Καλό σας απόγευμα, συνάδελφοι. Καθίστε. Και ας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας που προβλέπεται μέχρι τις 6.30 σήμερα το απόγευμα. Θα προεδρεύσω μέχρι να έρθει ο πρόεδρος. Το πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης και έχω μία πρόταση. Πρόταση αναβολής του σημείου 8, την έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ε, έκθεση αξιολόγηση σχετικά με την οδηγία ε, κράτησης δεδομένων. Και το θέμα αυτό θα αντικατασταθεί από μία δήλωση του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων του κυρίου Μανσερβίση σχετικά με την καινούργια ανακοίνωση της Κομισιόν που αφορά την εισρωή μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική και την ενίσχυση του Frontex και του μηχανισμού της Schengen. Αυτό αντικαθιστά το τωρινό σημείο 8. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη, οι αντιρρήσεις δεν βλέπω, δεν υπάρχουν σήμερα το απόγευμα ανακοινώσει του Προέδρου. Οπότε προχωρούμε στο σημείο 3. Εντολή για τον διάλογο, τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012. Συνάδελφοι, θα αρχίσουμε σήμερα με μια παρουσίαση από την Κομισιόν του Σχεδίου Προϋπολογισμού του 2012 που δημοσιεύτηκε στις 20 Απριλίου στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η Κομισιόν προτείνει αύξηση 17,7% στις υποχρεώσεις και 6,8% στις πληρωμές. Αυξήσεις είναι αυτές σε σύγκριση με το 2011. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την πρότασή τους και μετά θα λάβει το λόγο η συγγήτριά μας, η κυρία Κέλλερ, για να παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής της για το, την εντολή για το δημοσιονομικό τριμερή διάλογο του Ιουνίου που στοχεύει στον καθορισμό προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη του τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό και μετά θα κάνουμε ένα γύρο συζητήσεων. Οπότε πρώτα ο λόγος στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια. Ευχαριστώ και τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που δίνουν στην Κομισιόν την ευκαιρία να παρουσιάσει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012. Προτείνω να κάνω μια γενική παρουσίαση της πρότασης, υπογραμμίζοντας σε σημαντικά θέματα κυρίως. Όταν τελειώσω την παρουσίαση, ευχαρίστως να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Γενικό σχόλιο καταρχήν. Η προετοιμασία του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2012 έγινε στα πλαίσια των μικρών, ε, των ανωτάτων ορίων και της μηδενικής ανάπτυξης των ε, ε, ανθρώπινων πόρων για να λάβουμε υπόψη τα οικονομικά προβλήματα στα κράτη-μέλη. Ειδικότερα, το ύψος των ε, πιστώσεων πληρωμών εξετάστηκε και παρέμεινε σε ένα ελάχιστο όριο στο σχέδιο της Κομισιόν. Η παρουσίασή μου θα επικεντρωθεί στο 3α, ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, που είναι το 1% του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2012 από την Κομισιόν. Με άλλα λόγια, η κατηγορία 3α είναι 1,3 δις ευρώ από σύνολο 142 δις ευρώ. Παρά το δύσκολο οικονομικό πλαίσιο, η κατηγορία ότι το κεφάλαιο του Α βλέπει σημαντική αύξηση επιστώσεων υποχρεώσεων σε σύγκριση με το 2011, 17,7% συγκεκριμένα. Αυτό είναι 1,3 δις ευρώ. Αυτό αντικατοπτρίζει την πολιτική σημασία στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά την συνεχιζόμενη εξάπλωση του προγράμματος της Στοκχόλμης. Οι πιστώσεις ε, πληρωμών επίση αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο, το 2011 δηλαδή, κατά 6,8% και έτσι έχουμε σύνολο 868 εκατομμύρια ευρώ για λόγους σύγκρισης, σημαντικό αυτό, 17, το 17,7% και το 6,8% οι αυξήσεις δηλαδή αντίστοιχα για υποχρεώσεις και πληρωμές στο κεφάλαιο 3α θα πρέπει να ειδωθούν στο φως των αυξήσεων που είναι μόνο 3,7% στις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων και 4,9 πιστώσεις πληρωμών στο σύνολο του σχεδίου προϋπολογισμού της Κομισιόν. Το 3α λοιπόν θεωρεί αντιμετωπίστηκε ως προτεραιότητα με πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση από ό,τι είναι ο κανόνας. Δύο λόγια τώρα για το περιθώριο. Θυμάστε ότι είναι η διαφορά μεταξύ των συνολικών ποσών που έχουν ε, ε, ε, δεσμευτεί και την, στην δημοσιονομική περίοδο 2007-2013 και το ε, η πρόταση είναι για τον προπολογισμό του 2012. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό περιθώριο αν υπάρξουν απρόβλεπτα όπως η τωρινή κρίση στη Βόρεια Αφρική για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε ε, πρόσθετα κεφάλαια όποτε αυτά θα χρειάζονται. Το τωρινό περιθώριο του 3α είναι 65,6 εκατομμύρια ευρώ που είναι πάνω από το ενδεικτικό περιθώριο που κοινοποιήθηκε στη Δημοσιονομική Αρχή τον Ιανουάριο του 2011. Η αύξηση κατά 39 εκατομμύρια σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιανουαρίου προέρχεται από χαμηλότερο προϋπολογισμό για τον οργανισμό των συστημάτων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας. Τώρα, λεπτομέρειες. Γιατί τέτοια αύξηση για το 3α το 2012 αφού έχουμε την τωρινή οικονομική κρίση. Ουσιαστικά η αύξηση αντικατοπτρίζει την πολιτική σημασία του χώρου δικαιοσύνη και εσωτερικών. Συγκεκριμένα οι περισσότερες μεγάλες αυξήσεις συνδέονται με τα κεφάλαια ε, για την πολιτική αλληλεγγύης και διαχείρισης των ε, μεταναστευτικών ροών, solid funds πάγια και ολοκλήρωση, ε, ενσωμάτωση ε, υπηκών τρίτων χωρών κλπ. Αν τα δούμε τώρα αυτά, το κάθε ένα χωριστά, οι πιστώσει ε, για το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων είναι περίπου κατά 38%, πιστώσεις 16% σε σχέση με τις πληρωμές, αύξηση Οπότε έχουμε αύξηση 95 εκατομμύρια ευρώ στις πιστώσει υποχρεώσεων και 27 εκατομμύρια ευρώ για τις πληρωμές. Το 2012 προβλέπεται ότι θα χρηματοδοτηθούν νέες εξελίξεις σε πέντε τομείς στρατηγικής σημασίας που είναι προτεραιότητα για την Ένωση. Πρώτον, ε, έλεγχος της συμβατότητας συστημάτων με τα ε, προγράμματα ε, Schengen Information System το 2 επίσης η εξάπλωση του Visa Information System το VIS σε σημεία διασυνοριακά επίσης πιο σημαντική εφαρμογή του Visa Code που ισχύει από τον Απρίλιο του 2010 4. Η εισαγωγή εθνικών κέντρων συντονισμού και ανάπτυξη συστημάτων ώστε τα ευρωπαϊκά ε, σύνορα να τα εποπτεύουμε αποτελεσματικότερα το 2015 και να είναι λειτουργικό το νέο σύστημα και ε, τα παρόντα βέλτιστα στις ε, τεχνολογίες ελέγχου στα σύνορα όπως το έλεγχος στα σύνορα που είναι το γνωστό σύστημα, τα συστήματα μάλλον ABC. Δεύτερον, οι πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την ε, ενσωμάτωση υπηκών τρίτων χωρών αυξήθηκε κατά 23% για τις υποχρεώσεις και 5,1% για τις πληρωμές. Αυτό σημαίνει αύξηση 31, κατά 31 εκατομμύρια ευρώ για τις υποχρεώσεις και 4 εκατομμύρια ευρώ για τις πληρωμές σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011. Έτσι, Αυτές οι αυξήσεις αντικατοπτρίζουν τη σημασία και τις προκλήσεις του νέου Ταμείου Αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά τους νόμιμους μετανάστες εγκατεστημένους στο έδαφος της Ένωσης. Το Ταμείο θα συμβάλλει στην ε, εφαρμογή εθνικών στρατηγικών ε, ενσωμάτωσης υπηκόντρων τρίτων χωρών. Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας ενσωμάτωσης κάθε χρόνο. Το 2012 η αύξηση για την επαγγελματική κατάρτιση ε, για άλλα προγράμματα αγωγής πολίτη αυξήθηκαν για να διευκολυνθεί η πλήρης ενσωμάτωση των υπηκόντρων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, οι πιστώσεις που προτείνονται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών αυξήθηκε κατά 33% για τις υποχρεώσεις και 8,6% για τις πληρωμές σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 49 εκατομμύρια ευρώ στις υποχρεώσεις και 6 εκατομμύρια ευρώ στις πληρωμές. Κάτω το 2012 θα, το Ταμείο θα στηρίξει τα κράτη-μέλη στην ολοκληρωμένη διαχείριση επιστροφών και επίσης θα προβλέψει ε, κοινέ δράσεις από τα κράτη-μέλη προωθώντας έτσι την ε, ομαδοποίηση των, ε, της πραγματογνωμοσύνης και θα έχουμε έτσι εξοικονόμηση στην αποτελεσματικότητα. Δεν υπάρχει αύξηση στις ε, πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Η πρόταση της Κομισιόν για το 2012 στηρίζεται σε αυτή την προϋπόθεση στις δημοσιονομικές προοπτικές. Το ποσό που προβλέπεται για το 2012 είναι λοιπόν το ίδιο όπως και το 2011. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι είναι παρόλα αυτά αύξηση 38%. 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο ποσοστό. Και άλλες αυξήσεις της πρότασης της Κομισιόν χρήζουν προσοχής το σύστημα VIS, VIS και η πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος οι πιστώσεις για αυτό το συγκεκριμένο 38,8 εκατομμυρία για το 2012 είναι αύξηση 83% για τις υποχρεώσεις και 44% για τις πληρωμές σε σύγκριση με τον προπολογισμό του 2011. Αύξηση λοιπόν 17,5% ε, εκατομμύρια για τις πληρωμές και 8,8 ε, για τις πληρωμές. Μετά την τελική αποδοχή του συστήματος στο πρώτο τρίμηνο του 2012, η ανάπτυξη συμπληρωματικών λειτουργιών θα καταστεί αναγκαία, δηλαδή τροποποιήσεις, τροπολογίες στο Visa Code που εγκρίθηκε όπως σας είπα πριν τον Απρίλιο του 2010 και την αποδοχή των δαχτυλικών αποτυπωμάτων για να αποκλείσουμε το FTE failure to enroll. Αύξηση λοιπόν για τις υποχρεώσεις εδώ 8% 9 εκατομμύρια ευρώ συγκεκριμένα, μειώνεται όμως κατά 10,6% στις πληρωμές. Ε, διαχρονικά μπορέσαμε καλύτερα να χαρτογραφήσουμε τη σχέση μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών ε, πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι οι ανάγκες για πληρωμές το 2012 είναι λιγότερες. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για να υπάρξουν δράσεις προτεραιότητες όπως καταπολέμηση της διαφθοράς, καταπολέμηση της εμπορίας, την πορνογραφία το, με τα παιδιά, το έγκλημα και η παράνομη χρήση του διαδικτύου. Τώρα, για τους οργανισμούς δικαιοσύνης και εσωτερικών. Το 2012 το 3α θα στηρίξει 8 οργανισμούς. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων είναι εξαίρεση όμως γιατί θα συνεχίσει να υποστηρίζεται από την κατηγορία 1α στα πλαίσια των τωρινών δημοσιονομικών προοπτικών. Δύο από αυτούς τους οργανισμούς είναι στην αρχική φάση ή είναι νεοδημιουργηθέντες. Ε, το γραφείο ΙΑΖΟ για την ε, στήριξη του ασύλου στη Μάλτα και επίσης ε, το Οργανισμός για την στήριξη μεγάλων προγραμμάτων πληροφορικής. Τα άλλα έχουν συνεχίσει, η Frontex, η Europol, το Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Σάιλπολ, του Eurojust και το Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών, η NCDDA. Για να έχουμε το επίπεδο επιδοτήσεων του προηγούμενου έτους, η Κομισιόν έλαβε υπόψη την, ε, το στάδιο των εξελίξεων του οργανισμού, για παράδειγμα να μην υπάρξουν άλλες προσλήψεις ή δημιουργία θέσεων εργασίας ε, ε, για τις, τους οργανισμούς που έχουν ήδη απογειωθεί εκτός και αν πρικοδοτηθούν περισσότερο και βέβαια έσοδα από το 2010, δηλαδή τα πλεονάσματα από το 2010. Ε, δεν θα υπάρξουν νέες θέσεις, δεν συμφωνήθηκαν δηλαδή στο πρόγραμμα εγκατάστασης με εξαίρεση εκείνων των οργανισμών που πήραν περισσότερες, ε, περισσότερα καθήκοντα ε, αναδιάρθρωση στην Eurojust και κάποιοι άλλοι. Οι πιστώσεις για το Frontex στηρίζονται στην τωρινή εντολή της Frontex, αυτή είναι η μόνη νομική βάση που έχουμε πάνω στην οποία μπορούμε να ε, στοιχειοθετήσουμε πρόταση, αλλά αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί αφού όταν εγκριθεί ο τροποποιητικός κανονισμός που τώρα ε, τον επεξεργάζονται. Συμπεραίνω λοιπόν, η προτινόμενη αύξηση για το 3α ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη είναι σημαντική αύξηση και αντικατοπτρίζει πλήρως την πολιτική σημασία αυτού του τομέα της πολιτικής. Όμως ε, θα πρέπει ε, να δούμε μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια τη σημαντική αυτή αύξηση. Ε, το 3α είναι λιγότερο από το 1% του σχεδίου προϋπολογισμού της Κομισιόν για το 2012. Οι προτινόμενες πιστώσεις υποχρεώσεων συνάδουν με το δημοσιονομικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε στις 28 Ιανουαρίου φέτος από τη Δημοσιονομική Αρχή και μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2011. Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών ε, εξετάστηκε πολύ προσεκτικά και περιεκόπη όπου χρειάστηκε από την Κομισιόν. Και σε αυτά τα πλαίσια μια υπενθύμηση, αν το ύψος των υποχρεώσεων είναι χαμηλό, των ε, πληρωμών, μπορεί η Κομισιόν να ενισχύσει κάποιες γραμμές του προϋπολογισμού μέσω του μηχανισμού του προϋπολογισμού, ούτως ώστε τα απαραίτητα κονδύλια να διατεθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε, ε, Είναι σημαντικό αυτό γιατί στο 3α είναι 64,7% 65% η πιστητώση υποχρεώσεων πληρωμών που είναι ο χαμηλότερος λόγος των άλλων σε σχέση με όλες τις άλλες κατηγορίες δαπανών στον προϋπολογισμό του 2012. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Συγγνώμη που παρουσίασα τόσα ποσοστά και νούμερα, αλλά αυτό είναι αναπόφευκτο όταν παρουσιάζουμε προϋπολογισμό και ελπίζω να μην σας μπέρδεψα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Εμείς ευχαριστούμε και την Επιτροπή γενικότερα για την παρουσίαση που έκανε της δημοσιονομικής κατάστασης για το 2012. επιστρέφω στην Προεδρία και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, εθελούσια καθυστέρηση, καθώς ερχόμουν από τη Μαδρίτη. Λοιπόν, άργησε να φτάσει το αεροπλάνο μου. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου λοιπόν στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας η οποία φυσικά ε, θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον μετά από αυτά που ακούσαμε σήμερα, μετά από τις επίσημες δηλώσεις του Προέδρου Ομπάμα σχετικά με την τύχη του αυτοαποκαλούμενου ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης ε, ε, ο οποίος εντοπίστηκε, στοχεύτηκε και φωνεύτηκε Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε η κυβέρνηση του κυρίου Ομπάμα σε, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης η οποία διαξήχθη τις τελευταίες 20 ώρες. Λοιπόν, περιμένουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση και τις εξηγήσει οι οποίες θα δοθούν για αυτές τις ιδιαίτερα σημαντικές ειδήσει σημαντικές ε, για την παγκόσμια προσπάθεια καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ιδιαίτερα των εκδηλώσεων της τρομοκρατίας που ε, αποτελούν θα έλεγα μια συνολική απειλή. Ξέρουμε ότι επιτίθενται παντού, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στο Μαρόκο. Τα περισσότερα θύματα τους είναι φυσικά ε, μουσουλμάνοι Ελπίζω λοιπόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης να επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στα πλαίσια του πρώτου θέματος που είμαι διάταξη, δίνοντας το λόγο στον εισηγητή, την εισηγήτρια μάλλον, την κυρία Φραντσέσκα Κέλλερ, η οποία θα παρουσιάσει την, τη γνωμοδότησή της. Επανέρχομαι λοιπόν στα του προϋπολογισμού, λέει η κυρία Κέλλερ. Η γνωμοδότηση αυτή αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο, δεν αφορά αριθμούς. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε αριθμούς, θέλουμε όμως να μεταφέρουμε τις προτεραιότητές μας και τα θέματα που θεωρούμε σημαντικά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ συνοπτικοί. Αυτά τα οποία έχω βάλει εγώ στην πρότασή μου είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία θα πρέπει να βασίζεται ο προϋπολογισμός, ιδιαίτερα στις προτεραιότητες των τομέα των ελευθεριών, όπως περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Στοχόλμης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ζούμε περίοδους οικονομικής κρίσης και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί έτσι ώστε τα χρήματα να αδαπανώνται σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουμε. Περαιτέρω, αναφερθήκαμε στις αυξήσεις τις οποίες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που επηρεάζουν την Επιτροπή μας και περιμένουμε φυσικά με ενδιαφέρον και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο πολιετές ε, πλαίσιο το οποίο αναμένεται. Περνώ σε αυτά τα οποία θέλουμε να εντάξουμε στον τριμερή διάλογο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρεί μονίμως τα προγράμματα με βάση την δυνατότητα να πετύχουν τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκαν και να αναφέρει τα αποτελέσματα αυτά στο Κοινοβούλιο. Αυτή θα πρέπει να είναι, πιστεύω, η βάση για τις δημοσιονομικές μας βάσεις τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο τον επόμενο χρόνο. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν πιστώσεις όχι μόνο ή όχι κυρίως στην προσπάθεια καταπολέμησης προβλημάτων όπως η παράνομη μετανάστευση, αλλά απαιτείται επίσης και πιστώσεις, απαιτούνται και πιστώσεις για την αποτελεσματική προστασία των μεταναστευτικών ροών. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική χρηματοδότηση για τις νέες αποστολές της συνθήκης και από το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Νομίζω επίσης ότι έχει σημασία να λάβουμε υπόψη μας τον διαχωρισμό της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Ελευθεριών σε δύο διαφορετικές διευθύνσεις γενικές, κάτι το οποίο θα έχει δημοσιονομικές συνέπειες. Αναθεωρείται, όπως ξέρετε, η εντολή Frontex και θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια του νέου προϋπολογισμού. Τέθηκε άλλωστε το θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα προγράμματα τα οποία δεν έχουν ακόμα νομική βάση δεν θα πρέπει ε, να τύχουν χρηματοδότησης και θα πρέπει να τεθούν οι θέσεις αυτές σε, ε, αποθεματικό. Για το ΣΥΣ2 ένα σημαντικό τμήμα θα πρέπει να τεθεί ε, σε αποθεματικό γιατί δεν είναι ακόμα λειτουργικό το ΣΥΣ2. Αυτά είναι λοιπόν τα οποία θα ήθελα να συζητήσουμε στον τριμερή διάλογο. Ελπίζω να συμφωνείτε. Εφόσον έχετε επιπλέον θέματα μπορείτε να κάνετε σχόλια ή να κάνετε επιπλέον συμπληρωματικές τροπολογίες. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών δεν είναι μακριά. Είναι η 5η Μαΐου, 12η Μεσημβρινή και η ψηφοφορία θα γίνει στο τέλος Μαΐου και γι' αυτό πρέπει να έχουμε τις προτάσεις σας το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ για την σύντομη παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Επιτροπής μας που περιλαμβάνονται στη δική σας γνωμοδότηση και που εκφράζουν τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε στις συζητήσεις. Υπάρχουν αρκετοί που έχουν ζητήσει ήδη τον λόγο. Αν υπάρχουν και άλλοι, Γκόνς. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια των σοσιαλιστών γύρω από το θέμα αυτό. Νομίζω ότι η αύξηση η οποία αναφέρθηκε ήταν προγραμματισμένη και είναι συμβατή με την, με την εμβέλεια και τη σημασία του τομέα αυτού. να μου επιτρέψετε να κάνω κάποια σχόλια για το Frontex. Επί τη βάση της τελευταίας εντολής δεν μπορούμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό. Αν αναθεωρήσουμε όμως τον κανονισμό του Frontex, τότε θα πρέπει να αλλάξει και ε, η χρηματοδότηση και οι πιστώσεις για το Frontex. Συμφωνούμε επίσης και με τις προτεραιότητες οι οποίες αναφέρθηκαν σχετικά με τη χρηματοδότηση του Frontex. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να καλύψει και άλλους τομείς, όπως τον τομέα της διεθνούς προστασίας των μεταναστών και όχι μόνο τον τομέα καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Και οι δύο αυτοί τομείς θα πρέπει να υπογραμμιστούν δεόντως. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα σχόλια οι αρμόδιες υπηρεσίες ε, φυσικά δεν λειτουργούν ακόμα και όπου αυτό συμβαίνει οι πιστώσεις οι οποίες προβλέπονται θα πρέπει να τεθούν σε αποθεματικό και το ίδιο ισχύει και ε, η πρόβλεψη πιστώσεων για το ΣΥΣ2. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα θέματα συμπληρωματικά που θα θέλαμε να προταθούν για πιλωτικά τις επόμενες ημέρες και να τα προσθέσουμε και να δούμε αν τα πιλωτικά αυτά προγράμματα αξίζουν χρηματοδότησης για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Γκόνς, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τις αναφερθήσεις προτεραιότητες όπως μας τις εξήγησε η συνάδελφος Κέλλερ. Βεβαίως και θεωρώ ότι παρά την θεσμενή οικονομική συγκυρία ταυτόχρονα έχουμε και κάποια ανθρωπιστική κρίση η οποία σοβεί όσον αφορά αυτές τις ε, μεγάλες μετακινήσεις ε, ε, προσώπων από την Λιβύη κυρίως. Μιλάμε για 450.000. Επομένως, με τίποτα δεν μπορεί να υποτιμήσει κανεί αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο είπε ω πατριώτα η Φρανσίσκα σε σχέση με το ζήτημα τη διεθνού και επικουρική προστασία. Τώρα. Αυτού του είδους το ταμείο, αυτή η πρόταση της Επιτροπής Μιλούμε για μια αύξηση 49 εκατομμυρίων και 6 εκατομμυρίων. συγγνώμη, 6, 6, 49 εκατομμύρια λέει ο μιλητής και άλλα 6. Και μιλάμε για αύξηση 43% και 3% αντίστοιχη αύξηση. Μιλούμε για κάποιο είδου πιστώσει πληρωμών και ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ω κίνηση, ω τάση, γιατί αυτό θα δώσει κάποια συνέχεια στην πολιτική. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το Ταμείο για τους ε, πρόσφυγες του 2012, ε, θα πρέπει η προκοδότηση να είναι σαν το 2011. Όμως, με όλο το σεβασμό προς την Κομισιόν, παρακαλώ να μην κάνει τέτοιου είδους συγκρίσεις όπως έκανε. Γιατί μας λέει η Κομισιόν ότι είναι το ίδιο αυτό το Ταμείο ε, των ε, η πρικοδότηση αυτή είναι ακριβώς ίδια, ενώ έχουμε 38% αύξηση σε σχέση με το 2007. Και τι γίνεται, με, και, ε, ε, ωραία. Το 1948 τι έγινε, η αύξηση του έγινε 100%. Μα τότε δεν, δεν υπήρχε. Κακό το αστείο είναι αυτό το οποίο μας λέει. Δεν είναι δυνατόν να μας λέει τέτοια πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ σε αυτή τη δική μας την... Ε, Τώρα μας λέει ότι έχουμε 38% παραπάνω το 2007, διότι αυτό το οποίο όντω ισχύει είναι ότι το Ταμείο των Προσφύγων για το 2012 θα έχει την ίδια πρικοδότηση με το 2011. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να μας διευκρινίσει η Κομισιόν. Ε, δεν μας είπε και πάρα πολλά τι γίνεται όσον αφορά αυτό το, αυτό το, το γραφείο ασύλου στη Μάλτα. Δεν μας είπε κανείς τους ελληνικά στοιχεία. Επομένως, η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ταμείο των Προσφύγων Νέου τίποτε άλλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρος. Εγώ ευχαριστώ κύριε Διαστεμέρα. Στο αγγλικά. Άλλος συνάδελφος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Θέλετε να υποβάλλετε κάποια ερώτηση, να προτείνετε κάτι, να σχολιάσετε κάτι σε σχέση με την κυρία Κέλλα, την εισηγήτρια. είναι αυτή η περιπτώση. Τότε πριν λάβει το λόγο σαν κύριε Κέλλη, να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τη Επιτροπή, τον κύριο ε, Μάρι. Κύριος Μωράν. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι έχω σημειώσει σωστά όλες τις ερωτήσει που υπευλήθησαν και θα προσπαθήσω μία-μία να τις απαντήσω. Εδώ τώρα ενώ ταυτόχρονα θα, θα, θα ψάχνω τα στοιχεία για τον προπολογισμό του του, του, του, του Ταμείου αναφέρθηκε για τη Frontex συμφωνώ 100% με τα όσα ελέγχθησαν οπότε όλα εξαρτώνται ε, για το πότε θα εγκριθεί η νομική βάση οπότε θα κάνουμε τροποποιητικό προπολογισμό ή επιστολή για τη χρήση του 2012 Άλλη παρατήρηση αφορούσε το κατά πόσο θα καλύψουμε τις ε, ανάγκες της ένταξης που όπως τόνισα στην ε, εισαγωγή μου έχουν αναλυφθεί κάποια διαδήματα, έχει γίνει επιπλέον πρικοδότηση και όλα αυτά καταδεικνύουν πόσο σημασία αποδίδουμε στην υπόθεση αυτή. Τώρα για το αποθεματικό. Ελπίζουμε ότι αυτή η υπηρεσία IT θα την έχει για τη χρήση του 2011 ή 2013 για το SIS2. Θα το δούμε στην πορεία. Όπως λέγαμε και, για, όπως λέγαμε ε, και στην έκθεση πρόοδου που υπευλήθη στο Κοινοβούλιο πέρσι το φθηνό πορτρό, αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Ε, βέβαια και ο Γενικός Διευθυντής θα έρθει σήμερα κιόλα. Ε, κάποια στιγμή για να το συζητήσετε εμείς έχουμε πάρα πολύ καλά επίγνωση του πόσο χρειάζεται να γίνεται ταχεία έγκαιρη ε, απόκριση, αντίδραση γι' αυτό και μιλούσαμε για το 2012 οπότε ήδη έχουν δεσμευτεί κάποια κονδύλια από τώρα από τώρα, από φέτος 2011 για το 2012 και έτσι θα βοηθήσουμε και τη Μάλτα και την Ιταλία να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή όλη την ζωή του κόσμου. Θα σα τα πει, θα ο κύριος Γενικός αργότερα σήμερα. Τώρα, για το Ιάσο, διαφορετική είναι η χρηματοδότηση, δεν αφορά το Ταμείο των Προσφύγων και όσον αφορά το 2012 προτείνονται 10 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε και έτσι αναγνωρίζουμε ότι μόλις τώρα ξεκινά η πορεία της. Και από τα 2 εκατομμύρια πάμε στα 8 φέτος και άλλα 10 το 12. Οπότε και θα, θα είναι πλήρω ε, λειτουργική και θα μπορεί ακριβώ να λειτουργεί όπως είναι επιθυμητό. Τώρα όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις Όχι, όχι, δεν, δεν ήθελα να υποτιμήσω την νοημοσύνη σα όσον αφορά αυτό το Ταμείο Προσφυγών. Απλώ λέγαμε ότι έτσι όπω έχουν σήμερα οι προοπτικέ, οι δημοσιονομικέ, ε, για την περίοδο όπω είχαν τέλο πάντων 7 με 13, τα ποσά τα οποία έχουν διατεθεί για αυτό το σημαντικό ταμείο, σε αυτή τη φάση υπήρξε η αύξηση 38%. Όμω ξεκάθαρα εννοούμε ότι όσον αφορά το 11 σε σχέση με το 2012 δεν υπάρχει καμία αύξηση και παραμένουν σε 93,5 93,5 ε, εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, για να δευτερολογήσει η συγκεντριά μας, η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ για όλα όσα αναφέρατε. Συμφωνώ με Και γι' αυτό για να προσθέσω όλα αυτά να τα εντάξω στην έκθεση. Οπότε θα προσπαθήσω να προβώ σε έναν συντονισμό και να δούμε τι θα γίνει με τις ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Εμεί ευχαριστούμε. Αυτά όσον αφορά τη συζήτηση αυτού του ζητήματο. Οπότε τώρα να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Διότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών όσον αφορά το σχέδιο τη νομοδότηση είναι η 5η Μαου το μεσημέρι. 5 Μαου. 12 η ώρα. Η δε ψήφιση θα γίνει τον Μάιο στις 24 και 25. και η αντίστοιχη ψηφοφορία στην Επιτροπή των Προπολογισμών θα γίνει κατά τα μέσα Ιουνίου. Όπως πέρσι, η Επιτροπή των Προπολογισμών επίσης μας έχει ζητήσει να υποβάλουμε τις προτάσεις μας όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και έργα και τις προπροσκευαστικέ δράσεις, οπότε η σχετική καταληκτική ημερομηνία ε, θα οριστεί για τις 27 Μαΐου το μεσημέρι. Και θα ενημερωθείτε περαιτέρω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά. Και προχωρούμε στο επόμενο σημείο, το σημείο παριθμών 4. Αλλά πρώτα πρώτα σας ε, αναγγέλω ότι έχουμε το 4, μετά το 5 και μετά το 6, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο 6, το 6 είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε σας προειδοποιώ να έχετε έτοιμες να πάνε να βρείτε τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Όποιος δεν έχει, ας πάει να τα βρει να του τη στείλουν τέλο πάντων. Οπότε προχωρούμε στο σημείο 4. Συγκρότηση ενό μηχανισμού αξιολόγησης ούτω ώστε να αξιολογείται το κεκτημένο Σέγγεν. Η συγκητή είναι ο κύριο Κόλλη, ο οποίο πρόκειται να μα ε, να μας εξηγήσει σχετικά και τι έγινε ε, κατόπιν τη συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή μα Ιανουάριο και Μάρτιο. Πρώτα πρώτα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κόλλη τον εισηγητή κατόπιν να μα πει τι, τι πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου και κατόπιν θα λάβουν λόγο οι άλλοι συνάδελφοι. Διότι προσέχει ενδιαφέρον να ξέρουμε ποια είναι τα επιχειρήματα ε, μια που υπάρχει τώρα προστριβή μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπή όσον αφορά την επιλογή τη νομική βάση για αυτή την πρόταση, διότι από ό,τι φαίνεται ε, όλο και περισσότερο υπάρχει ρεύμα του να υιοθετηθεί το άρθρο 77 όσον αφορά την νομική βάση. Διότι έτσι δεν θα εμπλακεί το Κοινοβούλιο στην ε, λόγω διαδικασία. Άρα το 70 ή το 77. Θα μας τα πει ο κύριος Κόλλιο. Έχει το λόγο κύριε Κόλλιο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να σας πω ε, να σας πω το, πώς έχουν τα πράγματα, να σας πω ποιο είναι το θεσμικό πρόβλημα, διότι εμείς είχαμε απορρίψει την πρωτοβουλία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι είχαμε επικαλεστεί μια σειρά αιτιών ουσίας, αλλά και άλλος λόγος ήταν η νομική βάση. Η πρώτη τους πρόταση της Επιτροπής δεν μας προσέδιδε το δικαίωμα να εμπλακούμε στην απόφαση. Η κυρία Μάλστρομ, ευτυχώ, κατέβασε μια καινούργια πρόταση. Εκεί προεβλεπόταν συναπόφαση, όπου θα εμπλεκόταν το κοινοβούλιο. Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για μια σωστή κίνηση. Κατάλαβε η Επιτροπή ότι όταν συζητούμε για θέματα ασφάλειας Σέγγεν, θα πρέπει να εμπλέκονται όλα τα θεσμικά όργανα. Με ανησυχεί αυτή η πρωτοβουλία πέντε κρατών μελών. Γερμανίας, κάτω χωρών Φιλανδίας, Σλοβακίας και Σλοβενίας. Μου προκάλεσε απογοήτευση ότι και το Νομινό Βασίλειο και η Σουηδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ελλάδα. Μετά προσεχώρησαν επομένω. 13 από του 27 έχουν προσχωρήσει σε αυτή την επιλογή και πρεσβεύουν ότι θα πρέπει η νομική βάση να είναι αυτή που προαναφέρατε σωστά, το άρθρο 77. Επομένως, δεν θα λαμβάνεται υπόψη, δεν θα ακούγεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα εμπλέκεται. Διότι τα σενάρια είναι τα εξή. Πρώτον, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποσύρει αυτή την πρωτοβουλία, να κατεβάσει μια καινούρια. Και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Άλλο σενάριο είναι το Συμβούλιο να χρειάζεται ομοφωνία για να αλλάξει την ε, νομική βάση. Γιατί το παρόν 13 στους 27 δεν αρκούν. Όμως το ότι 13 από τους 27 προτίθενται να κάνουν τέτοια κίνηση, αυτό δεν είναι τα καλύτερα μαντάτα. Μια που ελπίζουμε σε κάποια αγαστή συνεργασία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου τόσο ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα καινούργιο σύστημα αξιολόγηση έγκαιρα. Χρειάζεται επομένω πρόεδρε αυτή η συνεργασία. Χρειάζεται ένα νέο σύστημα αξιολόγηση. Νέο μηχανισμό αξιολόγηση. έχει περισσότερο κοινωνικό χαρακτήρα, φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση και εμπλοκή των ε, θεσμικών οργάνων. Και να μην υπάρχει προσέγγιση και σύστημα διακυβερνητικό. Χρειάζεται ένα τέτοιο μηχανισμό να ε, τα περισσότερη διαφάνεια. Να Συμβουλή το Κοινοβούλιο για, για τον έλεγχο και για την απόδοση, για τη συνεργασία. Ένας μηχανισμός ο οποίος να έχει περισσότερη συνεργασία. Ναι. Την, υπάρχει σώρα συμμετοχή, επιτροπή κρατών μελών, όσον αφορά την πλήρη συμμετοχή και έτσι να μπορούν οι Ευρωπαίοι και οι εθνικοί εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν πλήρως. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να γίνεται καλύτερη χρήση των πόρων. Να συμμετάσχει το Frontex και να αξιοποιείται η εμπειρία και ανάλυση κινδύνου που έχει. Αποδοτικότερος μηχανισμός, μικρότερες ομάδες, λιγότερο βαριές. Και επίσης χρειαζόμαστε ο μηχανισμός αυτός να είναι πιο συνεπής. Με ακριβή αξιολόγηση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες και να προβλέπει κάποιους μηχανισμούς έγκαιρη διόρθωση και να μην υπάρχει πια η αίσθηση ατιμωρησίας. Όπως είπαμε και στην πρώτη λίγη απόψεων, εγώ είμαι κάθετα αντίθετος στο να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μην ισχύουν άλλο, μην ισχύουν άλλα για αυτούς που είναι στο Σέγγεν και άλλα για τους υποψήφιους προς ένταξη στο Σέγγεν. Και η αίσθησή μου από ό,τι έχω ακούσει εδώ πέρα ότι οι περισσότεροι εξημών συμφωνεί μαζί μου. Δεν θέλουν περισσότεροι εξημών δύο μέτρα και δύο σταθμά και γι' αυτό και δεν είμαι υπέρ του να έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, δύο διαφορετικές αξιολογήσεις όσον αφορά υποψήφιους και μέλη. Να ισχύουν για όλους τα ίδια. Όλοι να συμμορφώνονται στους ίδιους κανόνες και στα ίδια κριτήρια. Εγκατακλείδη κύριε Πρόεδρε. Να μην κάνουμε αυτό που κάναμε στο παρελθόν. Δηλαδή να εξετάζεται κατά πόσον κάποιος υποψήφιος συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν όταν πρόκειται να προσχωρήσει και μετά να παραμελούν να κάνουμε το ίδιο όταν μιλάμε για, την, το εσωτερικό της ε, Σέγγεν. Επομένω, θέλουμε ένα τέτοιο μηχανισμό ευρωπαϊκού ευρωπαϊκή προσέγγιση και να επιδέχεται, να είναι δυνατή να γίνει αξιολόγηση για μέλη, για υποψήφιου, κατά πόσον λοιπόν συμμορφώνονται με του κανόνε ε, τη συνθήκη. Και αν δεν συμμορφώνονται, να προβλέπεται και να εφαρμόζεται κάποιο μηχανισμό διορθωτικό. Εάν δεν, τα προβλήματα συνεχίζονται να προβλέπονται κυρώσεις. Δεν λέω ότι η έκθεσή μου είναι οριστική, διότι αποφασίσαμε να επιταχύνουμε για θεσμικούς λόγους την παρουσίασή της. Έχουμε πει αυτά στην αρχή. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δίνει τον εκτήριο λάκτισμα, τόσο ώστε να στείλει αυτό το μήνυμα προς το Συμβούλιο. Το ΔΕ Συμβούλιο Αύριο κιόλα θα συνεδριάσει σχετικώ, πολύ σημαντικό αυτό και εμεί γι' αυτό ήδη θέλαμε να το συζητήσουμε όσον αφορά τι ε, υπάρχουσε προτάσει. Επομένω δεν τείνουμε στάση αναμονή, ε, δουλεύουμε, επιταχύναμε τη διαδικασία για αυτό το λόγο. Ξέρω φυσικά και δεν είναι τέλεια, ε, τίποτα δεν είναι τέλεια, επιδέχεται διορθώσει η εκθεσή μου, όμω ελπίζω ότι με αυτή τη χρονική περίοδο του, του μηνό που προβλέπεται για τι τροπολογίε γιατί έτσι θα καθοριστεί ένας μήνας για του τροπολογίες. Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτόν τον μήνα περιθώριο θα μπορέσουμε να επιφέρουμε τις διορθώσει με τις τροπολογίε και έτσι να βελτιωθεί η έκθεσή μου. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να επιφέρουμε διορθώσεις ή στην έκθεση. Όμως Νομίζω ότι εδώ και τώρα πρέπει να γίνει αυτή η παρουσίαση για λόγους θεσμικούς όπως σας προανέφερα. Thank you for the work and for the presentation of the draft report. Now we... Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μοσχάγκα. Shakespeare. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Δεν είναι πολύ συχνό το να χειροκροτεί ο εισηγητής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Χαίρομαι λοιπόν που υποστηρίζει πλήρως τις προτάσεις μας. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεσή σας και οι οποίες θα ενισχύσουν το μηχανισμό και θα τον βελτιώσουν περαιτέρω έτσι ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα στη διάθεσή μας. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να τοποθετηθείτε στις μεμονωμένες τροπολογίες στη συγκεκριμένη φάση. Σχετικά τώρα, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σχετικά με τη νομική βάση να προτείνει ε, μια συγκεκριμένη πρόταση επί τη βάση του 77. Αλλά απ' την άλλη πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη νομική βάση η οποία προβλέπεται και από τη συναπόφαση και την πλήρη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ θα γίνουν νομίζω για το συγκεκριμένο θέμα περαιτέρω συζητήσει με το Συμβούλιο. Τώρα από τους προεδρεύοντες του Συμβουλίου, Γιάννος Τσατούρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι θα είμαι πάρα πολύ συνοπτικός, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Θα ήθελα να μπορέσω όμως να σας παρουσιάσω από πλευράς της Ουγγρικής Προεδρίας τις θέσεις μας γύρω από την κατάσταση της συζήτησης ε, στο συγκεκριμένο κανονισμό. Το σχέδιο αυτό του κανονισμού έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης από την αρμόδια Επιτροπή Σέγγεν του Συμβουλίου, την ομάδα εργασίας μάλλον Σέγγεν του Συμβουλίου, τρεις φορές μέχρι τώρα, τον μήνα Ιανουάριο εισαγωγικά έγινε μια εμβάθυνση της συζήτησης της περαιτέρω συζητήσει, συλλέγοντας ταυτόχρονα τις προτάσεις τις οποίες σταδιακά μας έκαναν τα κράτη-μέλη. Ένα τμήμα των κρατών μελών έχει θέσει ορισμένα ενιολογικά θέματα θα έλεγα ή να το πω καλύτερα ορισμένα στρατηγικά θέματα που συνδέονται με τις βασικές έννοιες του κανονισμού. Μπορούμε να γενικεύσουμε λίγο λέγοντας ότι τα κράτη-μέλη υποστήριξαν τις τάσεις οι οποίες προσπαθούν να καταστήσουν τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε πιο αποτελεσματικά. Σχετικά όμως με την κατανομή των αρμοδιοτήτων και σχετικά με άλλα επιμέρους θέματα, υπήρξαν αρκετές προτάσεις διαφοροποίησης και προτάσεις τροποποίησης. Γύρω από τα στρατηγικά, σαν παράδειγμα, θέματα, οι συζητήσεις συνδέονται με το θέμα της νομικής βάσης του μελλοντικού κανονισμού. Στον Απρίλιο ασχοληθήκαμε με, τον, με το θέμα της νομικής βάσης και ακούσαμε επίσης προσεκτικά και τις απόψεις της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου ένα μεγάλο τμήμα των κρατών μελών, όπως και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου, επιβεβαίωσαν ότι σχετικά με τη νομική βάση του κανονισμού θα ήταν προτιμότερο να επιλεγεί το άρθρο 70 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην χρησιμοποιηθεί το άρθρο 77 όπως κάποιοι είχαν υποστηρίξει. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, περιμένουμε ένα τελικό έγγραφο από πλευρά της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και ελπίζουμε επί τη βάση αυτής της γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και ελπίζω ότι την 30 Μαΐου όταν θα συνέλθει εκ νέου η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου θα τεθεί το θέμα εκ νέου και ελπίζω τότε να μπορέσουμε να έχουμε την τελική θέση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν δεν ξέρω ποιος έχει ζητήσει το λόγο, ποια μέλη θέλουν το λόγο για την παρουσίαση που έκανε ο κύριος Κοέλιο. Ο κύριος Εντσίου πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Κοέλιο για την έκθεσή του. Πρόκειται για μια πολύ ισόρροπη έκθεση η οποία θα έλεγα βελτιώνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς θέτει το θέμα των διπλών μέτρων και σταθμών σχετικά με τα μέλη, τα οποία είτε είναι μέλη της, ε, σε, του Σέγγεν είτε είναι υποψήφιοι για να ενταχθούν στο σύστημα Σέγγεν. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να αποφύγουμε περαιτέρω διακρίσεις, αρκετές έχουν υπάρξει μέχρι τώρα. Ελπίζω ότι θα πρέπει οι αρχές οι με την προστασία των, ευρωπαϊκών, των προσωπικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Οι αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχουν τεράστια εμπειρία στον τομέα αυτό και χαιρετίζω επίσης και την εισαγωγή ενός συγκεκριμένου άρθρου για την εμπλοκή του Frontex σε όλα τα κράτη-μέλη που έχουν πρόβλημα με την εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν. Το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης πρέπει να κυριαρχήσει. Οι χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρέπει να τύχουν βοήθεια και μέσω του Frontex, έτσι ώστε όλα τα κριτήρια του κεκτημένου Σέγγεν να γίνουν σεβαστά αυτή τη στιγμή βοηθηθούν οι χώρες αυτές και δεν μπορούν πάλι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε μόνο θα πρέπει να λαμβάνονται κυρώσεις εις βάρος τους. Σχετικά με την εισαγωγή νέων κριτηρίων για κύμανσης, όπως αυτό έχει τεθεί από τον κύριο Κοέλιο. Νομίζω ότι η απόφαση αυτή είναι μια σωστή απόφαση και θα πρέπει να γίνει δεκτή νέα κριτήρια όπως το ποσοστό διαφθοράς σαν παράδειγμα ή το επίπεδο του οργανωμένου εγκλήματος. Τέτοια κριτήρια είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθούν απτά. Είναι αδύνατο να υπολογίσει κανείς το επίπεδο διαφθοράς της ένα κράτος μέλος με αντικειμενικό τρόπο. Ένα άλλο θέμα το οποίο μου φαίνεται σημαντικό και το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί τουλάχιστον αναλυτικά στην έκθεση αφορά την αρχή της διαφάνειας. Θα ήθελα να καταθέσω μία τροπολογία προς την κατεύθυνση αυτή γιατί έχω την αίσθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις τις οποίες κάνουν οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Συμπερασματικά να πω ότι αυτός ο νέος μηχανισμός αξιολόγησης θα είναι ένα θετικό βήμα σε σχέση με τον παλαιότερο μηχανισμό. Θα διαχειριστούμε καλύτερα το χώρο Σέγγεν, δίδοντας την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν τις ευθύνες που έχουν αναλάβει. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα επίσης να εμπλέξουμε και το Frontex στη σύνολη διαδικασία. Για μια ακόμη φορά να κάνω μια συμπληρωματική παρατήρηση για την επιστολή που απίφθινε η Γαλλία και η Ιταλία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα τα προβλήματα τα οποία οδηγούν σε υπερβολικές κατασταλτικές δράσεις θα πρέπει να τα αποφύγουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπονομεύουμε και να θέτουμε σε αμφισβήτηση την ίδια την ύπαρξη του χώρου Σέγγεν. Η έκθεση Κοέλιο είναι αφεαυτής ιδιαιτέρως φιλόδοξη και δίδει λύσεις στα προβλήματα τα οποία περιλαμβάνονται στην Ιταλογαλλική επιστολή. Εάν τα κράτη-μέλη σαν παράδειγμα εμπλέκονται στις αξιολογήσεις οι οποίες γίνονται και αν η υπηρεσία Frontex αναλάβει τον ρόλο τον οποίο της αξίζει, ένα μεγαλύτερο δηλαδή ρόλο, τότε θα μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στην επιστολή των δύο χωρών. Συν της η δυνατότητα αποχώρησης από το χώρο Σέγγεν να είναι κάτι το ιδιαίτερος έκτακτο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δεχτούμε το κλέσιμο των συνόρων σαν μια συνηθισμένη πρακτική όποτε μια χώρα θεωρήσει ότι τη συμφέρει ή την βολεύει. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πίσω και η έκθεση αυτή δεν έχει σε καμία περίπτωση με την διαδικασία ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρωμανίας στο Σέγγεν η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από τέτοιες εξωτερικές παρεμβάσεις. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Βέμπερ θα ομιλήσω εκ μέρους της κυρίας Λάντφορτ που είναι η σκιώδης εισηγήτρια και συντονίστρια της Άλντε στην Επιτροπή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο για την έκθεσή του. Υποστηρίζουμε πλήρως την στάση την οποία κρατά στην έκθεσή του. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνολικής έκθεσης αυτό το οποίο προσπαθεί είναι να καταστήσει τη διαδικασία πιο αποτελεσματική, πιο αυστηρή αλλά και πιο διαφανή. Συμφωνούμε πλήρως λοιπόν με την ιδέα Τη αποφυγής με κάθε κόστος των διπλών μέτρων και σταθμών. Είναι απαράδεκτη και ε, δημιουργεί διακρίσεις. Είναι πολύ καλή η πρόταση την οποία κάνει ο κύριος Κοέλιο επίσης για την δυνατότητα συμμετοχής εν μέρη και του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας στην διαδικασία αυτή έτσι ώστε να μπορέσουν και οι χώρες αυτές να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους σε επίπεδο αστυνομικής συνεργασίας και προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ένωσης. Σχετικά με το θέμα της νομικής βάσης. Από ό,τι φαίνεται, οι συζητήσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζονται, ο πόλεμος ανάμεσα στα δύο όργανα συνεχίζεται, δεν βλέπω το τέλος του, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις φοβούνται τους πολίτες τους τόσο πολύ και τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο πολύ. Πολιτικά δηλαδή, όχι μόνο σε επίπεδο ε, θα έλεγα νομικό, δυσκολεύομαι να το κατανοήσω αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σαφές ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διαδικασία της συναπόφασης, είναι η κανονική, τακτική διαδικασία και θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να εμείνουμε στη νομική βάση την οποία αυτή προτείνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτά, αυτό είναι το μήνυμα νομίζω που πρέπει να παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. κύριος Έλτσεφ. Δεν έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Σέλτσεφ, όχι. Κυρία Στανόκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα. Μετά από αυτά που ακούσαμε. Φαίνεται ότι θα υπάρξει ευρεία συνένεση των περισσότερων τουλάχιστον πολιτικών ομάδων και εμείς οι πράσινοι συμφωνούμε με τον κύριο Κοέλιο είναι μια ισχυρή αυτή η στεναρή γραμμή λεύσης. Συμφωνούμε για το θέμα της νομικής βάσης και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Εμείς θα ψηφίσουμε και υπέρ της προσχώρησης Βουλγαρίας. Ε, έχουμε ψηφίσει. Ε, Γερμανίας. Θα θα ψηφίσουμε να μπουν στο χώρο Σέγγεν, αλλά είχαμε πει ήδη ότι είμαστε κατά των δύο μέτρων και των δύο σταθμών και σε σχέση με τη Ρουμανία-Βουλγαρία τα είχαμε πει αυτά και θα είμαι ευτυχής να το επαναλάβω μαζί με τους συναδέλφους αυτό ως δήλωση πάλι. Ωραία. Η κυρία Γιώτοβα. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Κολλιό για αυτό το σχέδιο έκθεσης όσον αφορά τον νέο μηχανισμό της αξιολόγηση για τον χώρο Σέγγεν και ε, να δούμε τι θα γίνει με όλες τις χώρες αυτές που ε, είναι, είναι μέλη και συμφωνώ με τον κύριο Κοέλιο ότι θα πρέπει τα ίδια κριτήρια να ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη. Να μην έχουμε μια κατάσταση δύο μέτρων και δύο σταθμών. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την ευθύνη αυτής της αξιολόγησης, οπότε και θα πρέπει πιο γρήγορα από τα πέντε χρόνια να στείλει τους εμπειρογνώμονες και αυτοί να αξιολογούν το τι ισχύει και να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ε, που ισχύει από σήμερα. Τώρα θέλουμε να υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις και ελπίζουμε να λάβουμε απαντήσεις. Πρώτον, η ανακοίνωση της Επιτροπής παραμένει επίκαιρη. Χρειάζεται ένα νέος μηχανισμός για αξιολόγηση της εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν. Και πρόκειται να μας προσθέσει αποτέλεσμα των ενεργειών τη Οικομισιόν στο άμεσο μέλλον. Τι μεταβολές βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να επιφέρουμε σε λίγο πρόκειται να ε, ψηφιστεί η προσχώρηση Βουλγαρίας-Ρουμανίας στο Σέγγεν. Πώς συνδέεται αυτή η προσχώρηση με τον μηχανισμό αξιολόγησης. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την επιστολή της περισμένης εβδομάδος. Και εκεί ο Δανός συνάδελφος ζητεί να μην υποστηριχθεί η προσχώρηση Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Θα πρέπει επομένως να γίνει πιο ολοκληρωμένη συγκεκριμένη συζήτηση για το θέμα αυτό. Οπότε τώρα γιατί και ένα γενικότερο θέμα. Αυτός ο μηχανισμός για την αξιολόγηση που θα υπάρξει, πώς θα λειτουργήσει εάν κάθε φορά απορρίπτουμε τα καινούργια κριτήρια. Εάν θεωρείτε ότι τα τεχνικά κριτήρια πληρούνται από αυτέ τι δύο χώρε, αυτό σημαίνει ότι αυτέ οι δύο χώρε είναι έτοιμε για προσχώρηση στο χώρο Σέγγεν. Ακριβώς όπως έγινε και με την προηγούμενη διεύρυνση του χώρου Σέγγεν. Τα ίδια κριτήρια ίου. Αλλιώς πάμε σε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γι' αυτό και ελπίζω ότι θα εγκρίνουμε κάποιους κανόνες που θα ισχύσουν ε, ισότητα για όλα τα κράτη-μέλη. Και εμείς ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων θα δώσουμε τις εγγύησεις που χρειάζονται όλα τα κρατή-μέλη και γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία να μπορέσει να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία τη συναπόφαση για να μπορέσουμε να έχουμε έναν άρτιο μηχανισμό εύρεθμα να λειτουργεί και να βοηθάει την ασφαλεία στην Ευρώπη. Έχουμε τώρα αυτή την κρίση με του πρόσφυγε και κανένα δεν θέλει να έχουμε Ευρώπη διότι τίτλο ω προ αυτό. Να είμαστε κατηγορηματικοί στο μήνα που θα στείλουμε. Θα πρέπει αυτοί που προσχωρούν στο, στο χώρο να προσχωρούν όταν πληρούν τα τεχνικά κριτήρια. Και ο μόνος λόγος για αναβολή προσχώρησης να είναι μόνο πολιτικός. Πολιτικός λόγος που βέβαια θα πρέπει να δικαιολογείται από το Συμβούλιο όταν τον επικαλείται και αν επομένως το Συμβούλιο θεωρεί ότι τα τεχνικά κριτήρια δεν πληρούνται και ότι θέλει να ανεβάσει τον πύχη, τότε θα πρέπει το Συμβούλιο να το πει συγκεκριμένα. Ποτέ όμως δεν θα πρέπει να αναμειγνύουμε τον νέο, τη νέα αξιολόγηση και την άλλη μεριά το θέμα της προσχώρησης της Βουλγαρίας Ρουμανίας. Ευχαριστούμε κύριε Γιώτοβα. Κύριος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω καλυφθεί από τους συναδέλφους στα περισσότερα θέματα. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ για τον κύριο Κοέλιο, τον εισηγητή μας, για την πολύ ισορροπημένη ε, για το ισορροπημένο σχέδιο της εισήγησής του. Να προσθέσω μόνο όσα είπε σχετικά με τα πέντε ε, κράτη-μέλη που ε, γίναν μετά 13, ότι η ανησυχία αυτή για το Σέγγεν, όπως εκφράστηκε και την περασμένη εβδομάδα από τη Γαλλία και την Ιταλία, ακριβώς για αυτούς τους λόγους εμείς έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να αξιολογήσουμε αποτελεσματικά, να προχωρήσουμε σε αυτά που προτείνουμε και να επιλύσουμε τα νομικά και τα τεχνικά ζητήματα προκειμένου να αρθούν αυτές οι ανησυχίες του μέλλον. Είναι σίγουρο ότι στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσουμε και άλλες πιέσεις και γι' αυτό ακριβώς οφείλουμε το κεκτημένο του Σέγγεν να το περιφρουρήσουμε και να το ενισχύσουμε με κάθε τρόπο. Και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να μην έχει λόγο το κοινοβουλίο μας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Η κυρία Νέντελ Τσέβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα όμως να ζητήσω να μου πείτε, να μου εξηγήσετε γιατί δεν έχουμε μετάφραση προς τα βουλγαρικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε διερμηνία προς τα βουλγαρικά. Οπότε και εμείς έτσι ε, επίσης δεν μπορούμε να μιλήσουμε και να εφαρμόσουμε στη γλώσσα μας. Η γλώσσα μας είναι ισότιμη με όλες τις άλλες. Πέραν αυτό. Θα πρέπει να συγχαρώ τον κύριο Κοέλιο για την έκθεσή του. Ξέρω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτό το οποίο ανέλαβε να κάνει, οπότε θα πρέπει έτσι να δούμε πώ θα βελτιώσουμε και με τι Κομισιόν και νομίζω επίση ότι θα πρέπει να δούμε τι εγγύσει εύρυθμη λειτουργία θα υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να ενημερώσουμε κάποιο τρόπο, να επικαιροποιήσουμε το κείμενο και επίση έχω να σα πω τρία τεινά συγκεκριμένα ε, για την έκθεση. Αλλά πρώτα, σα επισύρω την προσοχή στον κίνδυνο ο οποίο ε, υπάρχει όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση. Πάρα πολλές φορές όσον αφορά για Βουλγαρία και Ρουμανία έχουμε ε, ε, συσχέτιση αυτού του θέματος με άλλα. Και αυτό θα ήθελα να το πω ενώπιον όλων, ότι οι κανόνες αξιολόγησης τους οποίους σήμερα συζητούμε δεν πρέπει να οδηγήσουν σε επιπλέον κριτήρια, επιπλέον απαιτήσει από αυτές τις δύο χώρες για την προσχώρησή τους. Διότι συζητούμε τώρα για κάποια κριτήρια τα οποία να ισχύσουν για όλους όμως αυτά τα κριτήρια να μην έχουν ε, ως αποτέλεσμα την τροχοπέδη στην προσχώρηση αυτών των δύο χωρών. Επίσης, ε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει όντως κλίμα αμοιβίας εμπιστοσύνη. Έτσι θα λειτουργήσει καλά ε, ο χώρος Σέγγεν. Επίσης, είναι σημαντικό να έχουμε εγγυήσεις λειτουργίας του συστήματος επί τη βάση κανόνων κοινών για όλους. Ακριβώς όπως είπαμε να έχουμε τέτοια αμοιβή εμπιστοσύνη και αυτή η εμπιστοσύνη θα πιάσει τόπο αν έχουμε τέτοιου είδους κοινά κριτήρια. Κοινή αξιολόγηση για όλους. Οπότε δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον κύριο Κοέλιο με τις τροπολογίες 5 και 18 όσον αφορά το τι γίνεται όσον αφορά το ότι μια χώρα δεν μπορεί μόνη να διαχειριστεί μια κατάσταση και επίσης όσον αφορά τις διατάξεις για τις κυρώσεις είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα ούτως ώστε να διασκεδαστεί πάσα αμφιβολία όσον αφορά ε, την επικράτηση δύο μέτρων και δύο σταθμών. Οπότε συμφωνώ με τα όσα είπε ο εισηγητή ότι θα πρέπει να έχουν ίδια μεταχείριση όλα τα κράτη. Επίση, όσον αφορά τη λειτουργία και την συγκρότηση των αξιολογητών, των ομάδων αξιολογητών, θα πρέπει να δούμε το πώ θα μπορούν η δουλειά του να πιάσει τόπο και επομένω να ξεκαθαριστεί η εντολή γιατί Είπαμε Europol, Eurojust θα έχουν τις ε, ομάδες τους. Να δούμε τι εντολή θα έχουν αυτές οι ομάδες και να δούμε ακριβώς με ποιες υπηρεσίες πρόκειται να υπάρξει συνεργασία. Τι εμπειρογνώμονες πρόκειται να αποσταλούν από αυτές τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η Όλαφ τι ρόλο θα παίξει. Και άπαξ και μιλούμε για τέτοιου είδους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, τότε δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το σκοπό μας. Να μην έχουμε επικαλύψεις, να μην έχουμε διασπάθηση των πόρων και ακριβώς να μην μπλέκεται το ένα στα χωράφια του άλλου. Οπότε νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κείμενο πρόκειται να ε, έχουμε καλύτερη αποδοχή των αποφάσεων που θα ληφθούν και επίσης θα υπάρχει αμοιβιότητα τελευταία να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη διαφθορά, τι θα γίνει με το οργανωμένο έγκλημα. Όλοι θέλουμε να έχουμε ε, κάποιου είδους μέτρα που να καταπονημούν αυτό το φαινόμενο όμως είναι ένα φαινόμενο που πάρα πολύ δύσκολα αποτιμάται και αξιολογείται ε, είναι θέμα κοινή γνώμης το, το, ειδικό βάρος των φαινομένων αυτών άρα θα πρέπει και εμείς να ορίσουμε, να υιοθετήσουμε κάποια κριτήρια ξεκάθαρα, συγκεκριμένα και κατόπιν αυτά τα κριτήρια, αυτοί οι δείκτες αντικειμενικά να εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Σέγγεν και να δούμε αφού όταν μιλούμε για διαφθορά σε ποιους τομείς θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό και σε ποιο επίπεδο. Επομένως, να δούμε το ότι ε, κατά πόσον, αυτό το λέω για παράδειγμα, κατά, κατά πόσον το Σέγγεν θα πρέπει να ασχολείται με τη διαφθορά σε ένα μικρό δήμο ή κοινότητα μακριά από τα σύνορα της χώρας και κατά πόσο αυτό έχει να κάνει με την εθνική κυριαρχία, πόσο, πόσο αυτό μπλέκεται την εθνική κυριαρχία. Ε, και άλλη μια φορά, συμφωνώ με τον κύριο Κοέλιο Σας ευχαριστούμε κυρία Έλτσοβα Και όσον αφορά την, το, το, το ζήτημα της ε, διερμηνίας, από και προς τη βουλγαρική γλώσσα. Αυτό θα ληφθεί υπόψη, θα το σημειώσουμε και για την κυρία Γιώτοβα ισχύει κάτι τέτοιο. Euh, θα ληφθεί υπόψη και θα το ρυθμίσουμε. Για να δούμε τώρα, θέλουν άλλοι συνάδελφοι το λόγο. Εάν όχι, τότε θα δευτερολογήσει ο συγκεκριτής μας ο κύριος Κουέλιο διότι πρόκειται σαφώς από τη συζήτηση ότι έχει δημορφωθεί ευρεία συνένεση ή στην Επιτροπή μας. Όσον αφορά μια νομική βάση που θα εξασφαλίσει την πλήρη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με συναπόφαση. Άρα πρέπει να καταβληθεί πάσα προσπάθεια και να αποφύγουμε το να ισχύσουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Για το κατά πόσον γίνονται προσπάθειες τόσο ώστε να εφαρμόζονται και να σχήμα και να πληρούνται τα τεχνικά κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα όσα είπαν, για τα όσα ευγενικά είπαν και επίσης θέλω να ενθαρρύνω τους πάντες να κατεβάσουν τροπολογίες και έτσι να βελτιώσουν την εκθεσή μου. Έχουμε μπροστά μας ένα μήνα για να δουλέψουμε, για να το αυτό και επίσης ελπίζω ότι θα έχουμε πολλές τροπολογίες διότι είμαι βέβαιος ότι έχουμε ένα σωρό σημεία τα οποία επιδέχονται βελτίωση. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα των κυρώσεων. Είχε δίκιο ο συνάδελφος που το ανέφερε και έχουμε ένα σωρό σημεία στην έκθεσή μου. Οπότε και πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις. Είμαι σίγουρος για κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, πολλοί από όσο έλαβαν ε, το λόγο μας μίλησαν για τη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Γάλλου Πρόεδρου και του Ιταλού Πρωθυπουργού. Σε σχέση με αυτό σας αναφέρω ότι δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι θεμελιώδεις διατάξεις της συνθήκης του Σέγγεν. Το δε θέμα που ανέκυψε με Γαλλία και Ιταλία δεν ήταν θέμα που είχε να κάνει με τις διατάξεις αυτές. Ήταν θέμα εφαρμογής αυτό Όμως εμείς εδώ τι είμαστε, είμαστε ένα κοινοβούλιο και η αναθεώρηση της συνθήκης προβλέπεται επί τη βάση της συναποφάσεως να γίνεται. Εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, τότε να προχωρήσουμε στην συζήτηση. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες συγκεκριμένες προτάσεις για να αναθεώρηση, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα. Τέτοιου πολιτικά πυροτεχνήματα για αυτή την συνάντηση των δύο αρχηγών κρατών. Όμως, αν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το ρόλο αυτών των δύο χωρών και του Σέγγεν, το θέμα είναι το αν υπάρχει ασφάλεια στο χώρο Σέγγεν. Κατά τη γνώμη μου η ασφάλεια εξαρτάται από δύο εργαλεία. Πρώτον, SIS 2 το σύστημα πληροφοριών Schengen είπαμε αυτό να προχωρήσει το 2007 στο 2011 θα πρέπει να δούμε πως θα γίνουμε πιο αποδοτικοί να δούμε τι προστιμένη αξία υπάρχει όσον αφορά ε, από το SIS 2 σύστημα, το SIS 1. Επομένω, χρειάζεται ένα καινούριο σύστημα και χρειάζεται ένα σύστημα αξιολόγηση άλλο εργαλείο. Αυτό δηλαδή που τώρα συζητούμε να φτιάξουμε, κατά τη γνώμη μου, με αυτά τα δύο εργαλεία, με το SIS 2 και με το νέο σύστημα αξιολόγησης Schengen, μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια του χώρου Schengen. Έτσι και όχι με άλλου είδους αποφάσεις. Τέλος, Πρόεδρε. Θέλω να σας αναφέρω ότι με εκπλήσει η πρωτοβουλία αυτών των πέντε. Των πέντε και των άλλων που τους υποστηρίζουν ή στο Συμβούλιο. Των πέντε κρατών μελών. Πέντε συν οκτώ των δεκατριών από τους 27. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν καταλαβαίνω πώς το Συμβούλιο και τα δεκατρια αυτά κρατημέλη δεν πρόκειται να σεβαστούν το Ευρωκοινοβούλιο το οποίο είναι η φωνή των Ευρωπαίων. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό καν. Δεύτερον, δεν αντιλαμβάνομαι το πώς έχουμε όλα αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία επιθυμούν να αναθεωρηθούν αυτές οι διατάξεις και προτιμούν να επιλέξουν μια, μια βάση νομική που δεν επιτρέπει τέτοια αναθεώρηση. τρία. αυτό το 77 δεν δίνει το περιθώριο στο Συμβούλιο να θεωρήσει κάποιες, ε, κάποιες ε, διατάξεις. Ας πούμε, ε, συμφωνώ σε αυτό το σημείο που αναφέρθηκε για τις απροειδοποίητες επισκέψεις και τα άλλα που προβλέπονται χωρίς αλλαγή κριτηρίων, χωρίς κυρώσεις. Επομένως δεν νομίζω ότι υπάρχει συνέπεια λογική για αυτή τη φιλοδοξία των κρατών μελών να συγκροτήσουν ένα πιο αυστηρό, πιο αποδοτικό σύστημα. Από τη μια μεριά και από την άλλη να, να ζητούν νομική βάση που δεν βοηθάει. Ούτε καταλαβαίνω γιατί τα πρεσβεύει αυτά η Ιταλία που κάθισε εκεί προς το Συμβούλιο ότι ότι ε, συμφωνεί με το 70 και το 77 και μετά καθίσανε και με τον Σαρκοζή είπαν ότι θα πρέπει να αφιερωθούν οι κανόνε της συνθήκης του Σέγγεν. Ε, το να λέει κανείς ε, το ένα και μετά λέει το άλλο δεν κολλάει. Τώρα τελευταία παρατήρηση κύριε Πρόεδρε. Το ξέρετε και το ξέρουν και οι συναδελφοί μα ότι στο παρελθόν όλα τα θέματα για το Σέγγεν διεκπαιρεώθηκαν σε πρώτη ανάγνωση. Τα θεσμικά όργανα έκαναν τέτοιου είδους προσέγγιση. Και έτσι, συμφωνήσαμε, καταλήξαμε σε ένα κοινό κείμενο και επίσης κλείσαμε το θέμα στην πρώτη ανάγνωση. Αλλά για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει η προσέγγιση να είναι επικοδομητική, θετική από όλα τα θεσμικά όργανα. Όμως το Συμβούλιο τώρα δεν δημιουργεί το πιο δημιουργικό κλίμα για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό που θέλουμε και αν το Συμβούλιο αυτά τα 13 κράτη-μέλη θέλουν να μας αφαιρέσουν το, τη συμμετοχή στην συναπόφαση, ε τότε ίσως θα πρέπει να πάμε σε μια πλήρη διαδρομή και διαδικασία όλες τις αναγνώσεις. Αν κανείς θέλει να συνεργαστεί, θα πρέπει τότε να σέβεται τα θεσμικά όργανα. Το ΔΕ Συμβούλιο θα πρέπει να το καταλάβει αυτό. Υπάρχει παρεμβολή από κάποιο κινητό. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοέγιο. Ευρεία υποστήριξη νομίζω έχουν οι θέση σας. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο αυτής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τον μηχανισμό αξιολόγησης. Τέλος θα πρέπει να ανακοινώσουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών αποφασίστηκε να είναι η Τετάρτη 25 Μαΐου το μεσημέρι. Και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Λίμπε στα μέσα Ιουνίου, 15 και 16 Ιουνίου συγκεκριμένα. Ωραία. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, δηλαδή δικαίωμα ενημέρωση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, Έχουμε τη συνάδελφο Birgit Ζίπελ, την εισηγήτρια. Θυμίζω ότι η πρόταση οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το δεύτερο βήμα ενός ε, χάρτη πορείας για τα ε, διαδικαστικά δικαιώματα που εγκρίθηκε το 2009 από το Συμβούλιο και ε, ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ησυχία παρακαλώ. ησυχία. Ε, εφόσον θα μείνετε στην αίθουσα, παρακαλώ να ε, μην ομιλείτε και να παρακολουθείτε για να συνεχίσουμε. Το πρώτο βήμα αυτού του χάρτη πορείας ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την έγκριση της οδηγίας για τα δικαιώματα μετάφρασης και διερμηνίας σε ποινικέ διαδικασίες. Τώρα η εισηγήτριά μας, κυρία Ζίπελ, υπέβαλε το σχέδιο έκθεσής της στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στο τέλος του 2010, πέρσι. Και πάνω στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας προσανατολισμού που έλαβε χώρα στις 17 Μαρτίου φέτος πάνω σε αυτή τη βάση άρχισαν διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Έγιναν ε, τριμερείς ε, διάλογοι μέχρι τώρα και ε, έτσι έγινε μια πρώτη συζήτηση για όλο το κείμενο της προτινόμενης οδηγίας. Εμείς θα ακούσουμε από την κυρία Ζίπελ, την εισηγήτριά μας, την εισαγωγή, μετά θα δώσουμε το λόγο στην Ουγγρική Προεδρία, στον εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας και μετά θα κάνουμε μια συζήτηση. Κυρία Ζίπελ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, με αυτή την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν, η οποία έκανε μια ωραία παρουσίαση πρότασης οδηγίας και ευχαριστώ και τους εισηγητές που με τις τροπολογίες τους, τις προσθήκες τους που τις συζητήσαμε στην Επιτροπή συνέβαλαν και εκείνοι να δράσουμε προς το συμφέρον των πολιτών μας και να βρούμε μια πρόταση αποτελεσματική και λειτουργική. Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο μέχρι τώρα πρέπει να πω ότι διεξήχθησαν σε πολύ καλή ατμόσφαιρα, σε καλό κλίμα, ακόμα και αν ε, χρειάστηκαν κάποια θέματα να συζητηθούν περισσότερο. Ε, ελπίζω ότι στο μέλλον οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν επίσης να κινούνται μέσα σε ένα καλό κλίμα. Κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις πριν μπω σε ορισμένα σημαντικά θέματα των διαπραγματεύσεων. Στη... Ήδη από τον πρώτο τριμερή διάλογο είπαμε ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποβάλουμε στην Ολομέλεια προς ψήφιση ένα κείμενο αν στο κείμενο δεν περιλαμβάνονται οι λεγόμενοι πίνακες αντιστοίχησης, correlation tables. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Τα, οι πίνακες αυτοί πρέπει να ενσωματωθούν στην οδηγία ανεξάρτητα από τα άλλα θέματα που θεωρούμε επίσης ότι είναι μεγάλη σημασίας. Δεν θα επισέλθω σε όλα τα θέματα που συζητήσαμε μέχρι τώρα. Θα αναδείξω μόνο τα πιο σημαντικά θέματα, όπως σε όλες τις οδηγίες σχεδόν. Στο ποινικό δίκαιο υπάρχουν κάποια θέματα γλωσσικής φύσεως που πρέπει να τα διευκρινίσουμε και να δούμε κάποιες έννοιες, πώς χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν επίσης διαφορετικές απόψεις σχετικά με το εύρος της αναφοράς σε άλλα νομικά συστήματα, σε σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή σε ποιο βαθμό πρέπει ή δεν πρέπει να γίνεται η αναφορά, η αναφορα η μηνυα τους. Στις τεχνικές συναντήσεις θα βρουν μια κοινή λύση, πάντως είμαι πολύ αισιόδοξη. Επίσης υπάρχουν κάποιες ενοιολογικές δυσκολίες προκειμένου περί, περί του πεδίου εφαρμογής των μηχανισμών και του πεδίου εφαρμογή των δικαιωμάτων, του εύρου των δικαιωμάτων, γιατί δεν εναρμονίζονται τα επιμέρους δικαιϊκά συστήματα, αλλά όποιος ε, ενέχεται σε κάποια ποινική διαδικασία έχει κάποια δικαιώματα που του υποβάλλονται γραπτός. Και μαζί με το Συμβούλιο έχουμε δύο ε, διαφορετικές απόψεις. Εμείς ως Κοινοβούλιο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αποφασίσαμε ότι θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να παίρνει ο κατηγορούμενος όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες, όσο γίνεται πιο νωρίς και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τα παρέχουν όλα αυτά έγκαιρα και νωρίς τη διαδικασία γραπτός. Και έχουμε και ένα κατάλογο των δικαιωμάτων που πρέπει να αναφέρονται και που εμεί το διευρύναμε, φαίνεται ότι για το Συμβούλιο είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ενώ ε, εμεί στο Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε γιατί στα περισσότερα κράτη-μέλη τα δικαιώματα αυτά είναι δεδομένα. Πολλά δικαιώματα θα τα ε, επεξεργαστεί περισσότερο ο χάρτης πορεία. και πιστεύουμε ότι όχι μόνο δεν βλάπτει, αλλά αντίθετα βοηθεί να ενημερώνονται οι κατηγορούμενοι για τα δικαιώματα που μπορούν να έχουν και στο μέλλον μάλιστα, ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουμε στην περαιτέρω διαδικασία του χάρτη πορείας. Θα πρέπει δηλαδή και σε εθνικό επίπεδο να είναι γνωστό ποια είναι τα δικαιώματα αυτά. Βέβαια, κάποιος ο οποίος κατηγορείται ή είναι, θεωρείται ύποπτος θα πρέπει να ενημερωθεί και για την κατηγορία. Αυτό ε, είναι πολύ σημαντικό, όπως το δικαίωμα σιωπής. Θα πρέπει να γνωρίζουμε γιατί κατηγορείται, ποια είναι η υποψία που τον βαρύνει. Ε, εκεί χρειάζεται πληροφόρηση, ενημέρωση. Το συζητήσαμε το Συμβούλιο, όπως και το θέμα κάποιων αλλαγών και τροποποιήσεων που ε, λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του κατηγορητηρίου μετά από την έκβαση των ερευνών, που και αυτές πρέπει να ε, είναι γνωστές. Ένα άλλο επίμαχο θέμα, ένα θέμα προσυζήτηση είναι όχι μόνο ο τρόπος της πρόσβασης στο υλικό, στο αποδεικτικό υλικό που υπάρχει, αλλά περισσότερο επίσης το θέμα των εξαιρέσεων ε, σε ποιο βαθμό κάποια αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να, ενδεχομένως να μην δοθούν στον κατηγορούμενο. Εμείς ως ε, Κοινοβούλιο είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια ε, νομική απόφαση ως βάση και οι εξαιρέσει πρέπει να είναι όσο γίνεται λιγότερες. Οι εξαιρέσει που προτείνει το Συμβούλιο πιστεύουμε εμείς ότι είναι πολύ πιο ευρύτερες αλλά και πιο γενικά διατυπωμένες και σίγουρα εδώ θα χρειαστεί να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Άλλα θέματα προς συζήτηση, δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες, είναι το θέμα της εκπαίδευσης των συνεργατών μας, ούτω ώστε τα δικαιώματα αυτά να μπορούν να εφαρμόζονται αποτελεσματικά όπως και το ζήτημα περαιτέρω διευκρινήσεων, επεξηγήσεων ε, όταν είναι ε, ε, νοητικά καθυστερημένοι κατηγορούμενοι. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια επιστολή με τα δικαιώματα και με διευκρινήσεις. Επίσης, στη... έχουμε τώρα στις 11 Μαΐου και στις 30 Μαΐου τους επόμενους τριμερείς διαλόγους και θα δούμε τα επίμαχα θέματα και σε ποιο βαθμό μπορούμε να τα λύσουμε στα πλαίσια αυτών των δύο επομένων τριμερών διαλόγων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζίπελ, για την παρουσίαση αυτή. Για να δούμε τώρα από την Κομισιόν. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν θέλει να λάβει το λόγο. Η κυρία Κάρολαϊν Μόργαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Θα είμαι συντομότατη. Σύμφωνο με αυτά που είπε ο κύριος Ζίπελ, εμείς στην Κομισιόν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το επικοδομητικό πνεύμα και των τριών μερών στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Είναι καλές οι διαπραγματεύσεις, πολύ επικοδομητικό το κλίμα και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε επί ενός κειμένου μετά από δύο ακόμη τριμερείς διαλόγους. Είμαστε αισιόδοξοι για την επίτευξη της συμφωνίας. Ε, συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με το Κοινοβούλιο, σχεδόν σε όλα τα σημεία που έχουν μέχρι τώρα συζητηθεί, οπότε ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να δείξουν πνεύμα συμβιβαστικό, ούτως ώστε ε, σε κάποιο σημείο να συναντηθούμε. Ευχαριστώ. Και από την Προεδρία... Όχι, όχι ουδέν σχόλιον. Τότε τα δίνουμε το λόγο στα μέλη μας. Ο κύριος Αντωνέσκου. Η κυρία Αντωνέσκου, συγγνώμη. Με, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. ο πρόεδρος η κυρία Αντωνέσκου. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια. 14 θέματα συζητήθηκαν στους ε, ε, τριμερείς διαλόγους και υπήρχαν και υπάρχουν βέβαια και διάφορες έννοιες που θα πρέπει να φωτιστούν καλύτερα. Αυτό μένει να γίνει και υπάρχει ένα περιεχόμενο πεντάρθρων. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου το Συμβούλιο κάνει πιο γενικόλεγες διατυπώσεις ε, επειδή υπάρχουν διαφορετικά, ε, διαφορετικές ενόμεστάξεις τάξεις με διαφορές υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφορές μεταξύ δικαιικών συστημάτων οπότε είναι ένα θέμα ε, ποια ποινική διαδικασία θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 4 που είναι η επιστολή που καταγράφει τα δικαιώματα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται στο άρθρο 4 θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτός, εγγράφους. Τώρα, για τους πίνακες αντιστοίχησης και αυτό είναι ζήτημα κύριο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συγγήτρια πολύ σωστά το υπογράμμισε αυτό κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου. Σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης, σχετικά με το γιατί κάποιος κατηγορήθηκε ή συνελήφθη και τα δικαιώματα πρόσβασης στη δικογραφία. Εκεί σε αυτά δεν υπήρξαν μέχρι τώρα δυσκολίες και νομίζω ότι αυτά θα λυθούν όλα στο ε, επόμενο τριμερή διάλογο. Ο κύριος Άλμπρεχτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτρια. Κάναμε ένα καλό βήμα μέχρι τώρα στον τριμερή διάλογο και είναι αισιόδοξες οι προοπτικές για το μέλλον. Θα ήθελα να πω ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να κάνει και άλλα βήματα, όχι να συναντηθούμε στη μέση, αλλά θα δούμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Εγώ τρία θέματα θεωρώ κύρια. Από την αρχή ήταν σημαντικό το θέμα της ε, σειράς και των προσαρμογών, δηλαδή στα πλαίσια του χάρτη πορείας θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτό το έγγραφο δικαιωμάτων να προσαρμόζεται με βάση τα δικαιώματα τα οποία ενδεχομένως θα εναρμονιστούν σε μετέπειτα φάσεις του χάρτη πορείας. Είναι σημαντικό ως Κοινοβούλιο λοιπόν να συνεχίσουμε να πιέζουμε για το θέμα αυτό, ούτως ώστε να μην επιλέξουμε μια άκαμπτη διατύπωση, αλλά μια που θα επιδέχεται αξιολογήσεις και προσαρμογές. Ένα δεύτερο θέμα που μου είναι σημαντικό είναι οι εξαιρέσεις που αναφέρθηκαν και από την κυρία Ζίπελ για την πρόσβαση στα έγγραφα. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ξεκάθαρα θεωρώ ότι οι εξαιρέσει στην πρόσβαση θα πρέπει να είναι διατυπωμένες πολύ περιοριστικά και μια εξαίρεση ας πούμε όπως προς το συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον δεν είναι ε, σωστή γιατί κάθε έτσι ανοίγει ο δρόμος για οποιαδήποτε εξαίρεση και κατάχρηση. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Με καθαρή διατύπωση. Πολύ σημαντικό είναι η άρνηση της αναφοράς στην ε, νομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει ο ορισμός που, κυρίως που θα επιλέξουμε και οι πληροφορίες που θα συμπεριλάβουμε στην οδηγία να προσανατολίζονται προς την ομολογία του ε, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ. Ε, οι παρεμβάσεις έδειξαν συμφωνία μεταξύ εισηγητών και μεταξύ εισηγητών και κομισιών άρα ενισχύεται η θέση μας στις μετέπειτα διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και συμφωνώ με αυτό που είπε στην αρχή η Κομισιόν. Ε, είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι ότι κινείται το Συμβούλιο και στις επόμενες ε, συζητήσει στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου που είναι άλλες δύο ε, και θα δοθούν λύσεις εκεί. Ωραία. Ο Πρόεδρος. That having been said... Κατόπιν όλων αυτών προχωρούμε. Προχωρούμε στο επόμενο. We should be ready to move on. Προχωρούμε. Επαναλαμβάνει ο πρόεδρο, Η το σημείο τη διάρκεια που αφορά την ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δύο ψηφοφορίε, αν δεν κάνω λάθο. Πρόκειται για το σημείο υπαριθμών 6 και το σημείο υπαριθμών 7. Το 6 αφορά αυτό το τόσο λεπτό, δύσκολο θέμα όσον αφορά την εφαρμογή του Schengen, του κεκτημένου Σέγγεν σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Η είναι ο κύριος ε, Κοέλιο. Θα ψηφίσουμε για αυτήν την ε, έκθεση του κύριου Κοέλιο που αφορά την ε, σχετική αποφάση του Συμβουλίου. Παναλαμβάνει ο πρόεδρος για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν εις Βουλγαρία και Ρουμανία. 12 Απριλίου είχαμε την πρώτη εξέταση του σχεδίου κειμένου και 14 Τετάρτου ήταν η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες. Οπότε και επ' αυτού θα ψηφίσουμε τώρα. First, we hear Mr. Πριν όμως αρχίσει η συνεργασία, η ψηφορία, συγγνώμη, έχω το λόγο κύριο Σκόλιο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα, σύντομα θέλω να σας πω ότι ευχαριστώ όλους για αυτές τις τροπολογίες και θέλω να σας πω ότι θα ήθελα οι τροπολογίες 2, 3 και 4 να απορριφθούν, να τις καταψηφίσουμε, διότι με αυτές τις τροπολογίες ε, σκοπείται η αναστολή της προσχώρησης αυτών των δύο ε, χωρών στο Σέγγιν. δηλαδή το ανάποδο από αυτό που θέλω εγώ. Ακριβώς όπως έχει διατυπωθεί είναι έτοιμε οι δύο χώρε να προσχωρήσουν. Η τοπολογία υπαριθμών 2 καταλαβαίνω που το πάει. Συμφωνώ με το σκοπό αυτή τη διατάξεω, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να πάει ε, στο κείμενο για τον νέο μηχανισμό αξιολόγηση που σήμερα συζητήσαμε και όχι σε αυτό το κείμενο το οποίο αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για την προσχώρηση Βουλγαρία και Ρουμανία. Και για αυτό και ζητώ οι συνάδελφοι να καταψηφίσουν τις τροπολογίες 2, 3 και 4, αλλά να επιψηφίσουν τη δική μου υπαριθμόν 1. Και σας ευχαριστώ. Καλά λέει ο Πρόεδρος. Οπότε και τώρα θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία υπαριθμόν 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Ναι περί της ε, τροπολογίας 2 πρόκειται περί προφορικής τροπολογίας ή όχι για να ξέρω ότι εννοούμε και ψηφίσουμε το ίδιο πράγμα ναι ναι ναι έχετε δίκιο εδώ σημειώνεται ως ε, παρατήρηση ότι πρόκειται περί προφορικής τροπολογίας νομίζω ότι έχετε αυτό το κείμενο σας έχει διανεμηθεί αυτό το κείμενο και λέει ότι πρόκειται για προφορική τροπολογία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει διατυπώνει τον προβληματισμό του για την διαφθορά κλπ. Και τονίζει ότι όλα τα κρατημέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα μέτρα τους όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία την οποία και ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά αποχές θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Θεωρώ ότι έχει απορριφθεί, αλλά τέλος πάντων στο επιβεβαιώσουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, μπορει απορριπτεται απορρίπτεται. 13-2. Πάμε τώρα στην επόμενη τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά Αποχές. απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Πέρας. 33, 4, 3. Κατά 33, 3. Τότε καμία αποχή συγχαρητήρια κύριε Κοέλιο. Moving to the... Προχωρούμε τώρα στην άλλη έκθεση της κυρίας Σερακιάνη. Όσον αφορά το σχέδιο ε, απόφασης του Συμβουλίου, την, την πρόταση ε, απόφασης όσον αφορά την συμφωνία με την Κροατία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρατήρησης για τα ναρκωτικά και την εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο της σύστασης. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, προσέξτε. Ψηφίζουμε τώρα την γνωμοδότηση της κυρίας Σερακιάνη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. 33 2. Χωρίς αποχές. Εγκρίνεται και αυτό το κείμενο πέρας ψηφοφορίας. Και προχωρούμε στο επιπλέον σημείο το οποίο περιλήφθη στην ημερησία διάταξη. It is a deliberation, a discussion on the statement by Director General Stefano Manservisi on the incoming commission communication. Συζήτηση με τον κύριο Μανσερβίζη όσον αφορά το τι θα γίνει με αυτές τις μεταναστευτικές ροές από Βόρεια Αφρική. Παρακαλώ προσέξτε. Ο κύριος Μανσερβίζη στις 5 προβλέπεται να λάβει το λόγο. Επομένως έχουμε ακόμα 15 λεπτά. Άρα θα κάνουμε διάλειμμα 15 λεπτών και σε 15 λεπτά ξαναρχίζουμε.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 Ευχαριστώ.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

Dear colleagues, Thank you for your attention. Λοιπόν, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Thank you. First and foremost, we Λοιπόν, να καλωσορίσουμε για μια ακόμη φορά στις εργασίες μας τον Στέφανο Μανσερβίζη. Ο Μανσερβίζη είναι Γενικός Διευθυντής, υπεύθυνος για τις εσωτερικές υποθέσεις. Το θέμα έχει συμπεριληφθεί στις εργασίες μας σήμερα για να μπορέσουμε να ακούσουμε πού βρίσκεται η ανακοίνωση την οποία προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ισροές της μεταναστευτικές από τη Βόρειο Αφρική, σχετικά με την ενέσχεση του Frontex και σχετικά με το μηχανισμό Schengen. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρετε, τη ζητήθηκε ήδη να υποβάλει στο επερχόμενο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της 12ης Μαΐου τις προτάσεις της και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης Ιουνίου να υποβάλει μια πλήρη στρατηγική σχετικά με τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών από τη Βόρεια Αφρική μετά την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Και όταν λέμε Βόρειο τμήμα της Αφρικής εννοούμε την νότια Μεσογειακή Λεκάνη, μια τόσο σημαντική περιοχή για την Ένωση. Η συνεισφορά αυτή της Επιτροπής ζητήθηκε και από τον Πρόεδρο Σαρκοζή και από τον Πρωθυπουργό Μπερλουσκόνη. Έγιναν αρκετά σχόλια για το θέμα αυτό τις τελευταίες ημέρες, τις διαβάσαμε στον τύπο και γι' αυτό τώρα θα ακούσουμε από τον κύριο Μανσερβίση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συζήτηση στην Επιτροπή, τις απόψεις της Επιτρόπου Μέλστρομ συγκεκριμένα, η οποία θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Τζάι τις επόμενες μέρες και μετά ελπίζω να υπάρξει χώρος για συζήτηση. Έχετε το λόγο κύριε Μανσερβίζη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Assessment of the situation, obviously uh, the Λοιπόν, <clears throat> δεν μπορώ να μπω σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε γιατί ξέρετε ότι επιφυλασσόμεθα για τη συνάντηση τη 12 η Μαΐου. Αλλά παρόλα αυτά ε, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές θα τι αναφέρω. Θα ήθελα καταρχάς να παρουσιάσω μια κατάσταση της συζήτησης ε, και της κατάστασης επιτόπου. Σε αυτή τη φάση υπάρχουν 650.000 ε, ε, που έχουν εγκαταλείψει τη Λιβύη. 250.000 από αυτούς έχουν πάει στην Αίγυπτο, άλλοι τόσοι έχουν πάει στην Τινησία. Πολλοί έχουν ε, οδηγηθεί πίσω στη χώρα τους από τους αριθμούς που προανέφερα. Άλλοι είναι απομονωμένοι στα πλαίσια μιας πολύ κρίσιμης κατάστασης στη Λιβύη. Σχετικά με αυτούς που ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να μιλήσουμε για 32.000 στην Ιταλία, 32.000 στην Ιταλία πρόσφυγες και 1.500 στη Μάλτα. Φυσικά βέβαια οι αριθμοί αυτοί αλλάζουν συνεχώς, αλλά βρισκόμαστε σε αυτό το, σε αυτό το επίπεδο θα έλεγα. στην Ιταλία η πλειοψηφία αποτελείται από την Ισίους. Η Τινήση ε, δείχνει ότι κάποιοι από αυτούς έχουν ζητήσει διεθνή προστασία ή έχουν καταθέσει αίτηση για άσυλο. Στη Μάλτα όλοι όμως, οι 1500, 1200, 1300, δεν ξέρουμε ακριβώς, έχουν ζητήσει διεθνή προστασία. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες γιατί εξαρτώμεθα από τις πληροφορίες που μας δίνει το συγκεκριμένο κράτος δεν είναι τόσο την Ίση, αλλά είναι από τη Σομαλία, την Ερυθρέα και την Αιθιοπία. Και από το Σουδάν επίσης, οι οποίοι ζητούν, επαναλαμβάνω, διεθνή προστασία. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία κυριαρχεί στην περιοχή. Βλέπουμε όμως ότι τις τελευταίες ημέρες, λόγω ακριβώς της χειροτέρευσης της κατάστασης στη Λιβύη, ιδιαίτερα στην δυτική πλευρά της Λιβύης, έχουν υπάρξει πολλές αναχωρήσεις προς την Ιταλία. Στη Λαμπεντούσα υπάρχουν ε, Αφρικανοί από την υποσαχαρική Αφρική, όχι μόνο από το Κέρας, αλλά και από χώρες όπως το Τσάδα. Δεν έχουμε αναλυτικές πληροφορίες για το αν έχουν ζητήσει διεθνή προστασία αλλά εν πάση περιπτώσει <clears throat> η κατάσταση αυτών των προσφύγων είναι διαφορετική από τους ε, Τινησίους οι οποίοι είχαν φτάσει στην Ιταλία μέχρι τώρα. Τη στιγμή που συζητάμε λοιπόν τις εξελίξεις της κατάστασης στη Λιβύη βλέπουμε ότι οι παράμετροι αλλάζουν συνεχώς όχι μόνο τακτικοί σε εισαγωγικά οικονομικοί μετανάστες αλλά και άλλοι άνθρωποι από διάφορες χώρες οι οποίοι θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στη Λιβύη. Και είναι πολυθεμητό αν θέλετε το να ζητήσουν ε, μια διεθνή μορφή προστασίας. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη αριθμή, αλλά υπάρχουν κατά προσέγγιση εκτιμήσεις όπως είπαμε και βλέπουμε και ποιες είναι οι τάσεις οι οποίες διαμορφώνονται μετά από τα στοιχεία τα οποία έχουμε αναλύσει για τους κινδύνους και τις εξελίξεις. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει οικονομικά μέσα, πρώτον για ανθρωπιστικούς λόγους, έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι ε, βρίσκονται στην Τινησία, στην Αίγυπτο και στην Νότια Λιβύη και για αυτούς οι οποίοι έχουν αποβιβαστεί ε, σε άλλες χώρες Έχουμε περίπου δεσμεύσει 100 εκατομμύρια ευρώ ε, εν τη ευρία ενία για ανθρωπιστικούς λόγους. Έχουμε δώσει επίσης και ε, βοήθεια σε διάφορα μέσα για την προσωρινή τους εγκατάσταση. Έχουμε θέσει μέσα στη διάθεση των δύο κρατών μελών που υφίστανται την πίεση, την Ιταλία και τη Μάλτα, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτές τις αφήξεις σε επίπεδο χωριστικότητας, υποδοχής, ε, επαναπροώθησης όπου αυτό είναι εφικτό και ε, στα πλαίσια γενικότητα της κατάστασης ε, στον τομέα της υγιεινής περισσότερο όπου αυτό είναι εφικτό. Οι αποστολές αυτές είναι εν εξελίξη, θεωρούνται χρήσιμες και από την Ιταλία και τη Μάλτα αν και η Μάλτα δεν συμμετέχει άμεσα, αλλά παρόλα αυτά παίζει το ρόλο της. Εμείς δίδουμε μέσα, πλοία, αεροπλάνα και όπως βλέπετε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει η επιτάχυνση της μεταρρύθμισης της νομικής βάσης του Frontex έτσι ώστε να καταστεί ικανότερο και να κάνει περισσότερα πράγματα, να αναλάβει περισσότερες δράσεις όπως τεχνική βοήθεια προς τους εταίρους μας τους τινησίους και να μπορέσει το Frontex να είναι εγκύτερα στα σύνορα της Τινησίας και να βοηθήσει την ακτοφυλακή της Τινησίας να διαχειριστεί τα θαλάσσια σύνορά της. Ένα άλλο θέμα είναι η αναζήτηση περαιτέρω πόρων που θα πρέπει να προσθεθούν στον προϋπολογισμό του Frontex έτσι ώστε να μπορεί να κινητοποιεί περισσότερα μέσα, να παίρνει περισσότερες μορφές η παρέμβαση της Frontex και να αναλαμβάνει περισσότερες αποστολές στα πλαίσια των συζητήσεων που ήδη γίνονται. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία είναι υποσυζήτηση. Τώρα στα πλαίσια της συζήτησης με την Αίγυπτο και με την Τινησία σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε διάλογο σε υψηλό ε, υπαλληλικό επίπεδο όπως έχει προετοιμαστεί πολιτικά από το Συμβούλιο Υπαργών και μάλιστα περιμένουμε στις Βρυξέλλες, περιμέναμε στις Βρυξέλλες τον Πρωθυπουργό της Τινησίας ακυρώθηκε η επίσκεψη αυτή για λόγους εσωτερικούς αλλά εν πάση περιπτώσει ο διάλογος σε διοικητικό επίπεδο συνεχίζεται προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τις αναπτυξιακές προσπάθειες της τινησιακής κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει το θέμα των μεταναστών, των ανέργων Θέλουμε να βοηθήσουμε να βελτιώσει τις δυνατότητες της η την και σε επίπεδο θα έλεγα αποκατάστασης των θεσμών και να βοηθήσουμε σε ιεσδήποτε δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν να υπάρξει σωστή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και συνεπώς των μετανασταυτικών ροών πώς θα φυλάσσονται τα σύνορα, πώς θα οργανώνονται οι πτήσεις επαναπρόθεσης, πώς θα υποδέχονται τους ανθρώπους οι οποίοι επαναπροωθούνται ε, στα πλαίσια μιας νέας κατάστασης. Θα τα συζητήσουμε επίσης και στα πλαίσια του Περιφερειακού Προγράμματος Προστασίας για τους ε, πρόσφυγες οι οποίοι αναζητούν διεθνή προστασία στην Τινησία και σε περιφερειακό επίπεδο και επίσης έχουμε ξεκινήσει μακροπρόθεσμο διάλογο για την κινητικότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Στα πλαίσια του διαλόγου αυτού θα δημιουργήσουμε μια εταιρική σχέση όπως είπαμε στα πλαίσια της κοινή ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας της Άστον για να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη κινητικότητα των κοινωτικών μέσων στην περιοχή. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Περιγράφεται εν μέρη και στην επιστολή την οποία έστειλε η Επίτροπο Μέλστρομ στο Συμβούλιο την 11η Απριλίου και προσπαθούμε όλα αυτά να τα μεταφράσουμε στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η ενεξελίξη κατάσταση και ποσοτικά και ποιοτικά επιτόπου και τι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε. Ένα δεύτερο συστατικό της ε, υποδιαμόρφωση κατάστασης είναι το έκτακτο συμβούλιο του μηνός Μαΐου, το οποίο θα προετοιμάσει τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν και τον Ιούνιο για την Νότια Μεσόγειο αλλά και γενικότερα για τα μεταναστευτικά στην Ευρώπη. Προετοιμάζουμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση η οποία θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία με μια πιο μια μακροπρόθεσμη λογική. Θα αντιμετωπίζουμε και το μακροπρόθεσμο παράγοντα όπου είναι σαφές ότι η μετανάστευση και η νόμιμη μετανάστευση σωστά διαχειρισμένη είναι ουσιαστική για την Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους και θα πρέπει αυτό να γίνει εφικτό στα ένα πλαίσιο σεβασμού των νόμων, σεβασμού των κανόνων. Σε ένα πλαίσιο δηλαδή αντιμετώπισης όχι μόνο της ανάγκης που υπάρχει για υποδοχή της μετανάστευσης, αλλά επίσης και σεβασμού των αρχών, σύμφωνα με τις οποίες τα σύνορά μας θα πρέπει να δούμε πώς θα καταστούν πιο, ε, θα έλεγα, εύκολα διαχειρίσιμα και πιο ασφαλή γιατί τα εξωτερικά αυτά σύνορα είναι εξωτερικά για έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Δεν θα πρέπει μόνο σε περιπτώσεις κρίσης να βλέπουμε πώς θα τα διαχειριστούμε καλύτερα. Μία προσπάθεια που κάνουμε λοιπόν είναι να υπάρξει ένα καλύτερο ποιοτικό στάνταρ διαχείρισης των εξωτερικών σύνορων, ανεξαρτήτως από τις διάφορες θέσεις, να υπάρξει ένα ποιοτικό ευρωπαϊκό επίπεδο και μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση η οποία να βασίζεται πολύ στο Frontex, όχι μόνο σαν επιχείρηση διάσωσης αλλά και προληπτικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την κοινή θα έλεγα αντίληψη διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Να εφαρμόσουμε τα μέτρα αυτά και να βελτιώνουμε τις πρωτοβουλίες ε, που έχουμε ξεκινήσει έτσι ώστε η περιοχή να καταστεί πιο ασφαλής και μέσω της βοήθειας ε, να δώσουμε βοήθεια για να ολοκληρωθεί η σωστή διαχείριση των συνόρων και να διευκολύνουμε το πέρασμα των συνόρων σε όσους το δικαιούνται, όχι μόνο το αντίθετο. Και ένα άλλο θέμα είναι το πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα και τον χώρο Σέγγεν. Χώρο Σέγγεν σημαίνει όπως έχει ήδη ακουστεί πολύ τελευταία και δεν θα ασχολιάσω αυτά που γράφει ο τύπος, αλλά η αντίληψή μας λέγει ότι ο χώρος στο Σέγγεν υποφέρει από πάρα πολύ κυβερνητισμό θα έλεγα. Εμείς δεν είμαστε εξοπλισμένοι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση με μηχανισμούς αντικειμενικούς, με μηχανισμούς οι οποίοι να λειτουργούν σε διάρκεια. Λαμβάνονται επιτόπου αποφάσεις. Θέλουμε λοιπόν εμείς να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης Schengen, το οποίο να βασίζεται σε μια πιο κοινοτική αντίληψη, να υποστηρίζεται σε φυσικά από τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα στα κρατημέλη και στη Frontex και να κάνουμε τη σωστή αξιολόγηση και σωστές προτάσεις για να καλύψουμε τις, τα προβλήματα που έχουμε, για να καλύψουμε τις αδυναμίες που έχουμε, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε προληπτικά. Ένα δεύτερο θέμα στο οποίο σκεφτόμαστε σε αυτή τη φάση είναι να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτών που κάναμε μέχρι τώρα και ίσως να αντικαταστήσουμε μέχρι τώρα τον παρόντα μηχανισμό μονομερούς διακοπής της ισχύω με έναν πολυμερή θα έλεγα μηχανισμό όπως ακριβώς λειτουργεί ο μηχανισμός αξιολόγησης που θα δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει σε μια τελευταία φάση μόνο την δυνατότητα επανεισδοχής των ελέγχων στα σύνορα στην περίπτωση όπου τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση, δεν είναι ικανά να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύνορα με κατάλληλο τρόπο ή δεν είναι διαθέσιμα να κάνουν ένα τέτοιο έλεγχο με επαρκή και κατάλληλο τρόπο. Λοιπόν, θέλουμε να περάσουμε από αυτή την πλήρη διακυβερνητική αντίληψη που ισχύει σήμερα σε μια κοινοτικότερη αντίληψη η οποία να βασίζεται στη σωστή αξιολόγηση που θα οδηγεί στην δυνατότητα να καταργούμε την ισχύ του Σέγγεν με πολύ περιορισμένο τρόπο στο τελευταίο στάδιο εν πάση περιπτώσει και όπου επιβεβαιούται η αδυναμία του κράτους μέλους. Λοιπόν αυτά για τη διαχείριση των συνόρων. Τώρα ένα δεύτερο πεδίο είναι <clears throat> αφορά την κίνηση των προσώπων αυτών στο εσωτερικό της περιοχής Σέγγεν. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη ενσωμάτωση των τακτικών μεταναστών έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά όλα τα προβλήματα τα οποία ξεκινούν με την άφηξη αυτών των μεταναστών στις διάφορες χώρες και να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε αυτά σε ένα καλύτερο πλαίσιο. Εδώ τίθεται και το θέμα της καλύτερης διαχείρισης του συστήματος βίζας. Το σύστημα μέχρι τώρα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που είπα συνολικότερα για το πεδίο Σέγγεν. Υπάρχουν θετικά, υπάρχουν αρνητικά. Είδαμε ότι πρόσφατα μετά από την απελευθέρωση των θεωρήσεων στα Βαλκάνια υπήρξαν εντάσεις λόγω της κατά, κατάχρησης του συστήματος αυτούς από ορισμένου εταίρους. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό παρακολούθησης, θέλουμε να βασίσουμε τους μηχανισμούς μας σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού. Θεωρούμε επίσης ότι είναι χρήσιμο να προτείνουμε ένα μηχανισμό ο οποίος στην περίπτωση πλήρους απελευθέρωσης του συστήματος θεωρήσεων, σε περίπτωση μαζικών αφήξεων, σε περίπτωση καταχρήσεων να υπάρχει ένας κοινοτικό μηχανισμός ο οποίος να διακόπτει την απελευθέρωση των θεωρήσεων για μια χώρα, ε, για μια χώρα η οποία ίσως να μην συνεργάζεται, να το πω κάπως τεχνικά, μια χώρα η οποία παρουσιάζει εν πάση περιπτώσει προβλήματα στις ε, κινήσεις των ατόμων όπου υπάρχει κατάχρηση αυτών οι οποίοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας παράνομα χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις, συζητούν καταχρηστικά άσυλο κτλ. Σταθμίζουμε λοιπόν από τη μία τις ελευθερίες με τους κυρωτικούς μηχανισμούς από την άλλη, εφόσον ορισμένες προϋποθέσεις ε, το απαιτούν. Επαναλαμβάνω ότι αυτό θα γίνεται πάντα υπό πλαίσιο μεταξύ των οποίων και τον δικό σας έλεγχο και μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα τρίτο πεδίο είναι το της ενίσχυσης της ανάγκης να καταλήξουμε σε συμφωνία για το κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου μέχρι το τέλος του 2012. Νομίζω ότι αυτό είναι τμήμα της εικόνας που έχουμε μπροστά μας, να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας έδωσε το Συμβούλιο τον Ιούνιο, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Θα καταθέσουμε τις αναθεωρισμένες προτάσεις μας στο τέλος Ιουνίου Ξέρουμε ποιες είναι οι προτάσεις που γίνονται για τον Τούρνταξ του Λονδίνου. Ελπίζουμε λοιπόν τον Ιούνιο να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις δυνατότητες για μια πιθανή λύση. Ξεκάθαρα λοιπόν λέμε στην ανακοίνωσή μας ότι το σύστημα χορήγησης ασύλου είναι ένας ξεκάθαρος πυλώνας του ευρωπαϊκού προτύπου διαχείρισης της μετανάστευσης και θα πρέπει να ξεκινήσουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που φροντίζει αυτούς που χρήζουν διεθνούς προστασίας και που προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα χώρο ο οποίος θα προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και θα δώσει άσυλο σε αυτούς που το δικαιούνται. Τίθεται βέβαια εδώ το θέμα του να προχωρήσουμε με τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για τις συμφωνίες επανεγκατάστασης Ξέρετε και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για μια ακόμη φορά ότι προσπαθούμε να ξεκινήσουμε εκ νέου μια δεύτερη φάση προγραμμάτων ιδιαίτερα για τη Μάλτα και προσπαθούμε παράλληλα έτσι ώστε να ξεμπλοκάρουμε κατά κάποιο τρόπο την πρόταση που είχαμε κάνει για την επανεγκατάσταση. Είχαμε επίσης συζητήσεις με τους αρμοδίους για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε έστω και για μία περίοδο χρονική η οποία ανακαλύπτεται από την παρούσα νομοθεσία και ε, προσπαθούμε να, να προχωρήσουμε και σε αλλαγές στην παρούσα νομοθεσία γνωρίζοντας ε, τα προβλήματα και τις δυσκολίες τις οποίες δημιουργούν οι επανεγκαταστάσεις αυτές. Πολλά λοιπόν ακούστηκαν και από εσά, πολλά από αυτά θα ανταλάβουμε υπόψη μας στις επόμενες προτάσεις μας και θα στείλουμε ένα μήνυμα νομίζω σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή το οποίο θα οδηγήσει στο ξεμπλοκάρισμα της κατάστασης. Ένα τελευταίο θέμα είναι θα έλεγα η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή στις βασικές αρχές μας μέχρι το τέλος του φθινοπόρου έτσι ώστε η εταιρική σχέση για την κινητικότητα και την ασφάλεια να καθοριστεί σαν μια γενική κοινοτική πολιτική, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα της κινητικότητας και της μετανάστευσης να είναι τμήμα της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην είναι κάτι το ξεχωριστό, να είναι ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής μας και ε, η πραγμάτωση αυτής της προσπάθειας θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες εκπλήρωσης των στόχων, επίτευξης μάλλον των στόχων που θέτουμε. Πιο συγκεκριμένα, σε μια τελευταία φάση θα προτείνουμε τη συγκεκριμένη εφαρμογή της αντίληψης αυτής στην νότια περιοχή της Μεσογείου με τις χώρες της Βορείου Αφρικής θα ξεκινήσουμε συζητήσεις με τις χώρες αυτές <clears throat> για να ορίσουμε καλύτερα τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε και να τις εντάξουμε θα έλεγα σε μια προσπάθεια διασφάλισης της σωστότερης διαχείρισης των συνόρων τους, ασφάλειας των δημοσίων εγγράφων τους και διαχείρισης της επανεγκατάστασης όλων των δυνατοτήτων που δίδονται επί τη βάση του υπάρχοντος κώδικα Σέγγεν, όπου πολλά γίνονται όπως ε, η κοινή ε, ε, υποβολή αίτηση για τη χορήγηση ασύλου, να αυξήσουμε τον αριθμό θεωρήσεων για πολλαπλές εισόδους, που όλα αυτά μπορούν να γίνουν με το υπάρχον σύστημα, Τεχνικά βέβαια όλα αυτά είναι εθνικές αρμοδιότητες, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα κλίμα όπου τα πράγματα να εξελιχθούν καλύτερα και να συμπεριλάβουμε λοιπόν περισσότερα χαρακτηριστικά κινητικότητας για ερευνητές, για φοιτητές, για όλους τους καλή τυπίστη ταξιδιώτες, επιχειρηματίες και να διευκολύνουμε επίσης και να προχωρήσουμε και σε μια περαιτέρω φάση, σε μια απελευθέρωση του συστήματος θεωρήσεων. Αυτό τώρα ακούγεται πολύ φιλελεύθερο, αλλά παρόλα αυτά, αν υπάρξει περισσότερη ασφάλεια, μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα για να δείξουμε ότι μετά από την αποκατάσταση των πραγμάτων και μετά από την εφαρμογή στόχων στα πλαίσια κοινών συμφερόντων, ιδιαίτερα για τους νέους επιχειρηματίες, φοιτητές κτλ, η κινητικότητα μεταξύ της Βόρειας Αφρικής και της Ένωσης μπορεί να βελτιωθεί πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η, η δομή της τάση την οποία θα υιοθετήσει επίσημα την Τετάρτη το σύνολο των Επιτρόπων. Θα είναι η βάση της συζήτησης του Συμβουλίου Τζάι της 12ης Μαΐου και ε, ακριβώς θα είναι και η βάση ε, για τη συζήτηση που θα γίνει στο Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό τον Ιούνιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δήλωση και για τις ε, προβλέψεις για την πορεία της ανακοίνωσης τις επόμενες μέρες. Τώρα θα κάνουμε συζήτηση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας γιατί έχουμε και ένα άλλο σημείο και κλεισμένων των θυρών. Ο κύριος Πρίμπε θα μας πει για το PNR, τα δεδομένα από τις καταστάσεις επιβατών. Οπότε μην ε, κάνουμε μεγάλες ε, τοποθετήσεις ε, τώρα προτείνω να έχουμε ένα γύρο των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Κοέγιο ίσως από το ΕΛΚ. Δεν έχω ερωτήσεις για να είμαι ειλικρινής. Τρία σύντομα σχόλια θέλω να κάνω, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Δεν χαίρομαι πολύ όταν ακούω για νέα συστήματα γιατί πρώτα πρέπει να ολοκληρώσουμε τα συστήματα που χρειάζονται όπως το ΣΥΣ2 και μετά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε καινούρια. Σημερίζομαι τη γνώμη σας για την ε, συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, αλλά χρειάζονται κάποιες, χρειάζεται κάποια προσοχή, ούτως ώστε η τοπική συνεργασία στα πλαίσια του Σέγγεν να γίνεται σωστά εμείς έχουμε έναν ε, ε, αξιωματικό ασφαλείας ε, που μπορεί να συνεργάζεται δίπλα σε έναν αξιωματικό από τρίτη χώρα και θα πρέπει να είναι η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά δεδομένα θα γίνεται μόνο από τους δικούς μας αξιωματικούς χωρίς διαρροές εμπιστευτικών δεδομένων προς τρίτες χώρες. Πολλά πρέπει να σκεφτούμε σε σχέση με αυτό το θέμα. Για να υπογραμμίσω λίγο αυτό που είπατε εσείς για το Σέγγεν και τα, τις κατεπίγουσες ανάγκες τους. Τι είναι το Σέγγεν, ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη κυκλοφορία. Και για πολλά μέλη του Κοινοβουλίου το ε, Σέγγεν είναι ένα από τα σύμβολα της Ευρώπης. Φοβάμαι λοιπόν όταν ε, αποδυναμώνουμε τα σύμβολά μας, γιατί μπορεί η Ευρώπη να αποδυναμώνεται από την χρηματοοικονομική κρίση, αλλά το Σέγγεν δεν πρέπει να αποδυναμωθεί. Φοβάμαι ότι καμιά φορά παίρνουμε αποφάσεις ή κάνουμε πολιτικές δηλώσεις που αποδυναμώνουν το χώρο Σέγγεν. Πρέπει να φροντίσουμε το σύστημα αυτό όταν κάποιος κάνει ας πούμε συνοριακούς ελέγχους με ένα σύστημα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή προσέγγιση. Καμιά φορά και η κοινότητα ολόκληρη πρέπει να κάνει το ίδιο. Αλλά αυτά θα πρέπει να τα συζητούμε στα πλαίσια των, του νέου μηχανισμού αξιολόγησης του Σέγγεν. Όχι έξω, δεν είναι άλλη απόφαση. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση και να ληφθεί η απόφαση στα πλαίσια του, συστήματο του συστήματος μηχανισμού αξιολόγησης. Κύριε κ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Είναι περίεργο να μιλάμε βράχη και μακροπρόθεσμα μέσα σε ε, την πολιτική μετανάστευση σε δευτερόλεπτα. Είναι μεγάλη η ανακοίνωση αυτή για τη μετανάστευση. Μιλάμε για το Σέγγεν, τη συνθήκη του Σέγγεν που είναι ιδρυτική, εμβληματική Επίση, προσωρινού μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε κατεπίγουσες καταστάσεις στη Μεσόγειο και μιλάμε επίσης και για την πολιτική μετανάστευση τη Ένωση, Σε εποχή λιτότητα, σε εποχή όπου όλοι αντιδρούν στεναρότατα κατά της μετανάστευσης. Και το πακέτο για το άσυλο επίσης, εις επίμετρον αυτό, που πρέπει να είναι έτοιμο το 2012. Διαβάζω από την επιστολή αυτή μετά τη, τη γαλλογερμανική. Θα έχουμε ένα σύστημα πριν από το 2012 με μόρφη ε, βιώσιμη. Τώρα ασκούνται ήδη μεγάλες πιέσεις σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια, η ερώτηση τώρα δεν είναι προς την Κομισιόν, αλλά στο Συμβούλιο. Υπάρχουν τόσες αντιφάσεις, τόσο βαθιές αντιφάσεις, που πραγματικά είναι σουρεαλιστική η κατάσταση θα πρέπει να καταπιαστούμε με θέματα που μπορούμε να λύσουμε και να διαχειριστούμε. Στην ανακοίνωση, και αυτή είναι ερώτηση αν θέλετε, ούτως ώστε να κάνουμε κάποια πρώτα. Ε, ρωτήσαμε για την προσωρινή προστασία την κυρία Μάλμστρομ, την οδηγία δηλαδή για προσωρινή προστασία και ρωτάμε γιατί δεν έχουμε σύστημα ασύλου έτοιμο ε, το οποίο θα επιμερίζει τις ευθύνες. Και είχαμε, συνέχεια καθυστερήσεις και τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στη Μεσόγειο. Αυτό είναι παλιό ε, αίτημα όχι μόνο ενός κόμματος. Τι θα λέτε για αυτά τα θέματα στην ανακοίνωση. Θα πείτε για παράδειγμα ότι πάλι δεν συγκεντρώνεται η πλειοψηφία η απαραίτητο στο Συμβούλιο, ότι η Κομισιόν θέλει να τεθεί σε εφαρμογή ο μηχανισμός. Αυτά είναι κάποιες θεματικές ενότητες που μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε... Είναι πολύ δύσκολο να πιάσουμε γενικόλογα όλο το θέμα, το ευρύτερο αυτό θέμα. Επίσης για το Σένιν, η εγγύηση που θέλουμε διαπαραταξιακά, όχι μόνο ένα κόμμα για το Σένιν, είναι ότι υπάρχουν μηχανισμοί για να γίνονται ας πούμε έλεγχοι στα σύνορα για λόγους δημόσιας τάξης. Και έχουμε και ένα διακυβερνητικό σύστημα, peer review. Αυτό θα κάνει, δηλαδή το peer review θα ε, παγιωθεί σε κάποιο μηχανισμό που να επιτρέπει τους ε, ελέγχους στα σύνορα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν και περισσότερα κράτη-μέλη και αυτά που δεν θίγονται άμεσα. Αυτά είναι κάποιες διασφαλίσεις που θέλουμε να υπάρχουν στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Ε, να, ε, δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα. Για το πακέτο του ασύλου και το πακέτο της μετανάστευσης που πάλι βρίσκει σύμφωνο τα κόμματα διαπαραταξιακά, τι θα γίνει στο Συμβούλιο. Είναι στενές, μικρές οι και θα έχουμε πρόβλημα τους επόμενους μήνες. Μπορεί η Κομισιό να συνεχίσει να λέει και να προσπαθεί και να λέει ότι όλα πάνε καλά. Και εμεί συμφωνούμε σε πολλά μέτρα μαζί σας. Το Συμβούλιο τι θα κάνει όμως και τι θα το κάνουμε. Μπορεί να είναι απλοϊκό το ερώτημα. Αλλά φαίνεται ότι και για, το, και για τα δύο πακέτα μετανάστευσης και ασύλου θα υπάρξει πρόβλημα στο Συμβούλιο γιατί έχουμε λιτότητα, υπάρχουν φόβοι στο Συμβούλιο. Οπότε τι θα κάνουμε. Όταν θα παρουσιάσετε την ανακοίνωση της Κομισιόν, πώς θα το κάνετε. Θα παρουσιάσετε τη θέση σας ως μια πραγματικότητα που θα επιδέχετε κάποιες πρόοδους, που θα δούμε πού. Γιατί φοβάμαι ότι θα κολλήσει το πακέτο για τη μετανάστευση, λόγω εξωτερικών παραγόντων επίσης. Όχι λόγω του έργου που επιτελεί η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριος Μούλντερ τώρα, παλαιό μέλος, από το Φιλελευθέρους. Ε, θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Εγώ διάβαζα την απόκριση, τα απάντηση του κυρίου Μπαρόζο στο, στη γαλλογερμανική επιστολή και απόρρισα λίγο. Ανεξάρτητα από το αν είναι κανείς υπέρ κατά του Σένιεν, Νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα είναι, είναι εφικτό να γίνονται έλεγχοι στα σύνορα πάλι στην Ευρώπη, αν γίνεται ας πούμε μεταξύ στα σύνορα τα γερμανοολλανδικά, θα έχετε μια συμφόρηση κυκλοφοριακή από το Άμστερνταμ μέχρι τα σύνορα την ώρα της εχμής. Λοιπόν, πώς βλέπει η Κομισιόν το ενδεχόμενο ε, πρακτικής εφαρμογής των ελέγχων στα σύνορα, όπως είπε ο κύριος ε, Μπαρόζο. Η κυρία Σαρτζεντίνη από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα σχέδιο μπροστά μου ε, της ανακοίνωσης για τη μετανάστευση και στη σελίδα 6 θα διαβάσω, από τη σελίδα 6 θα διαβάσω ένα απόσπασμα για την διακυβέρνηση Σέγγεν. Ένα μηχανισμό πρέπει να εισαχθεί και που θα επιτρέπει σύντονη και προσαρρινή επανεισαγωγή ελέγχων σε διάφορα σημεία των εσωτερικών συνόρων. Και λέει στο τέλο η Κομισιόν διερευνά την, τη φυκτότητα εισαγωγή τέτοιου μηχανισμού και μπορεί να υποβάλει σχετική πρόταση σύντομα. Και ρωτώ, τι είναι σύντομα, τι σημαίνει το σύντομα, πότε θα είναι, τι σημαίνει σύντονε, τι σημαίνει προσωρινός. Και το πολιτικό μου ερώτημα έχει ως εξής. Εσείς υποβάλατε προτάσεις για παράδειγμα για τους εποχικούς, τους ε, ICTs. Δεν προχωράει το θέμα στο Συμβούλιο αφού το Συμβούλιο δεν είναι πρόθυμο να ε, συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα για μετανάστες ένα πρόγραμμα για μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης κλπ. Πώς θα γίνει λοιπόν μετά από μια κρίση θα υποβληθεί πρόταση για ε, εσωτερικούς ελέγχους στα σύνορα χωρίς σαφή κριτήρια. Αν αυτά τα προβλέψει για την επόμενη Τετάρτη, ξέρετε ότι... Α, λέει ότι σύντομα θα υπάρξει πρόταση. Ε, μπορείτε να μας πείτε ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Ποιος άλλος θέλει να κάνει δήλωση ή ερωτήσεις. Δεν βλέπω. Η κυρία Ιντσφελτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορώ να σας τα πω πάρα πολύ γρήγορα και έχω κάτι για τα πρακτικά και μια ερώτηση. Η παρατήρηση είναι ότι με εντυπωσίασε το ότι η επιστολή για Γαλλία και Ιταλία απεστάλλει από τον πρόεδρο της Επιτροπής και όχι από τον υπεύθυνο, τον αρμόδιο επίτροπο. Αυτό για μένα έχει πολιτική σημασία. Η ερώτησή μου αφορά αυτήν την ε, προσωρινή ε, ε, καθιέρωση αυτών των ελέγχων. Αυτό το έχω υποβάλει ως κοινωνική ερώτηση και ξέρουμε τι γίνεται. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι δικαιολόγητο. Από την άλλη μεριά όμως, σε κάποια περίπτωση, αυτό έγινε επειδή ο Πάπας θα πήγαινε στην Μάλτα ή σε άλλη περίπτωση συνάντηση κορυφή στην Πορτογαλία και όταν ρωτούμε αν μπορεί η σε αλλη περιπτωση συναντησε κορυφη στην πορτογαλια και οταν ρωτουμε αν μπορει η πορτογαλια να μας εξηγήσει γιατί δικαιολογούνται αυτοί οι έλεγχοι λένε δεν μπορώ να πούμε γιατί αυτό είναι απόρριτο είναι θέμα εθνικής ασφάλειας οπότε με τίποτα δεν θεωρώ ότι αυτά είναι αποδοτικά και δεν θεωρώ εν τόσο ότι δικαιολογούνται αυτή η προσωρινή έλεγχη στα σύνορα. Ευχαριστώ. Εγώ λέει ο πρόεδρος και δίνω το λόγο στην κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ και εγώ συμφωνώ με αυτές τις αμφιβολίες που διατυπώθηκαν τους προλαλήσαντες και έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, είπαμε ότι θέλουμε έναν ε, μηχανισμό για ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί λοιπόν είπαμε, να κάνει τέτοιου είδους προτάσεις Κομισιόν σε συγκεκριμένε περιπτώσεις. Σε ποιες περιπτώσεις όμως προβλέπεται αυτή η αρμοδιότητα της Κομισιόν το κατεπήγον πώς ορίζεται, ποιος αποκρίνει εάν συντρέχει κατεπήγον ή ου και τι γίνεται με τα κράτη-μέλη εάν δεν συμφωνούν θα ξαναγκάζονται. Τι θα γίνει. Θα υπάρχουν από τη μία μεριά και όχι και από την άλλη των συνόρων ε, έλεγχος. Θα υπάρχει τοπικός περιορισμός. θα ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέρη. Δεν, δεν έχω καταλάβει. Επίση, τι γίνεται. Η, ο μηχανισμό που ισχύει σήμερα, ότι δηλαδή τα κράτη-μέλη μπορούν να κρίνουν ότι θα κάνουμε ελέγχου γιατί έρχεται ο Πάπα δεν ισχύει πια, δεν μπορούν να, να κάνουν κάτι τέτοιο. Επίσης, και όσον αφορά την κατάργηση των θεωρήσεων διαβατηρίων, θέλω να ρωτήσω το ίδιο. Ποιος κρίνει αν έχουν ε, έρθει πάρα πολύ, ας πούμε, σε μια χώρα και έτσι κόβει τις βίζες. Ευχαριστώ πολύ και τώρα κυρία Σίπελη, ο πρόεδρος, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αναρωτιέμαι γιατί μιλάμε τώρα για την ανανέωση του Σέγγεν. Αναρωτιέμαι δηλαδή για τα χρονοδιαγράμματα. Βλέπουμε έτσι ένα ρεσιτά λιθοποιίας των δύο αρχηγών κρατών Μπερλουσκόνη Σαρκοζή που κάνουν ως εάν η Ευρώπη είναι ανίκανη να ελέγξει τα σύνορά της με... και τώρα δημιουργούν μια τεχνητή κατάσταση που δεν τη θέλει κανείς γιατί δεν θέλουν να περνούν από την Ιταλία και να πηγαίνουν στη Γαλλία οι μετανάστες και θέλουν να συζητήσουν με τεχνητό τρόπο το θέμα των εσωτερικών ελέγχων στα σύνορα, στο έδαφος του Σέγγεν. θα μπορούσαν να αποσταλούν στην Τινησία αφού δεν ζητούν άσυλο. Γιατί πηγαίνουν στη Γαλλία, γιατί αποστέλλονται εκεί. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα του χώρου Σέγγεν, είναι πρόβλημα δύο αρχηγών κρατών που δεν είναι σε θέση ή δεν είναι πρόθυμοι αντικειμενικά να καταπιαστούν με το πρόβλημα και κάνουν αντιπερισπασμό ε, ε, επειδή θέλουν ε, χρήματα περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερα ακόμα άλλα. Σίγουρα εμείς ε, δεν ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στους πτυχιούχους και στους ε, υπηκόους τρίτων χωρών υψηλής ειδίκευσης. Ο στόχος είναι η ανειδίκευτοι. και τα προβλήματα δεν είναι τα κορυφαία στελέχη του management, είναι οι ανειδίκευτοι ή χαμηλής ειδίκευσης μετανάστες που έρχονται εδώ για να απασχοληθούν κάπου. Αυτό είναι κοινωνικό πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα του Σέγγεν, είναι θέμα διαμόρφωσης των αγορών εργασίας μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αυτά τα πλαίσια της υποκριτικής των Μπερλουσκόνη και Σαρκοζή, δεν έχει νόημα, είναι λάθος ε, η σηματοδότηση που θα ε, στείλουμε αν μιλήσουμε για διαφοροποίηση του Σέγγεν. Γιατί και προς τις τρίτες χώρες θέλουμε λάθος μήνυμα, αλλά και στους δικούς μας τους λαούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Μανσερβίζη, ακούσατε τις ερωτήσεις από τις πολιτικές ομάδες, από τους καθένα των βουλευτές της Επιτροπής μας. Αν μπορείτε να απαντήσετε. Μανσερβίζη. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που είπατε, τις επικρίσεις σας, ε, όλα αυτά και θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι προανέφερα ότι τον Απρίλιο το Συμβούλιο μας είπε να προβούμε σε κάποια ανακοίνωση. Βραχυπρόθεσμα αλλά και άλλη μία μακροπρόθεσμη. Επομένως η ανακοίνωση στην οποία θα προβούμε δεν τα καλύπτει όλα, δεν είναι ενδελεχής. Όμως στόχος μας είναι να καλύψουμε ένα σωρό πράγματα και ένα σωρό προβλήματα. Δεν θα βρείτε εγώ εκεί κάποια στοιχεία λεπτομέρεια. θα υπάρξει μια άλλη ανακοίνωση που θα εγκριθεί όταν ήρθε η ώρα. Άρα εκεί δεν θα βρείτε λεπτομέρειες. Ανακοίνωση που αφορά την ασκουμένη πολιτική. Για να δούμε πού πάει η μετανάστευση, διαχείριση συνόρων, ελεύθερη διακίνηση, τέτοια ζητήματα. πώ θα τοποθετούμε στα σχέση με του συνομιλητέ μα. Άρα δεν θα βρείτε λεπτομέρειε για τον μηχανισμό. Αυτό θα γίνει μετά. Αφού αποφανθεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αν συμφωνούν ή όχι. Επομένως, έχουμε μια τέτοια ανακοίνωση και θα ακολουθήσει η πιο μακρόπνοη. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε τη σύνοδο του Ιουνίου που θα το συζητήσει. Συγκεκριμένα πράγματα. Και ελπίζω ότι το Συμβούλιο πρόκειται να χαράξει κάποιες κατευθυντήριες, κάποιους προσανατολισμούς για το τι θα κάνουμε για το άσυλο. Επίσης όμως θα εγκρίνει και κάποιες γραμμές πολιτικής που θα ακολουθήσουμε. Να ποιος είναι ο στόχος αυτής της ανακοίνωσης. Και για πρώτη φορά προσπαθούμε να μην έχουμε κατάτμιση της πολιτικής, να έχουμε μία γραμμή όσον αφορά τη των συνόρων και έτσι όλοι κατά αυτόν τον τρόπο να μπορούν να κινούνται πιο άνετα. Τώρα, όσον αφορά πιο συγκεκριμένε ερωτήσει. Πρώτος ο κύριος Κόλλιο. Για να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα-πρώτα να κάτσουμε και να βασιστούμε στα όσα έχουμε πετύχει για να άρουμε κάποιες, ε, κάποια προβλήματα. Και τι να έχουμε, νομοθετική πρόταση ή να έχουμε ένα πολιτικό έγγραφο. και είπαμε ότι δεν αρκεί μια συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο. Να συμφωνεί, να δούμε πώς θα σταθμίσουμε τα αντιμαχόμενα συμφέροντα. Έχουμε κάποια τεχνικά θέματα και είπαμε αντί για πρόταση θα κάνουμε ανακοίνωση. Και μετά θα συζητήσουμε με συμβούλιο, με συμβούλιο και με κοινοβούλιο. Τώρα επίσης όσον αφορά την συνεργασία στο Σέγγεν αυτό αφορά τα κρατημέλη όχι τρίτες χώρες. Τοπική συνεργασία. Και να έχουμε εναρμόνιση του καθεστώτος χορηγήσης θεώρησης. Έτσι να δημορφωθεί μια συνένεση. Ας πούμε την πολλαπλή βίζα να βγήσουμε την τα έξοδα και την γραφειοκρατία. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στον κόσμο. Κοινό κέντρο υποβολή, ε, ειδήσεων. Μην πηγαίνουν ε, στην Άγκυρα όλοι οι Τούρκοι να έχουμε στον Καζιαντέπ, α πούμε. Όλα αυτά μελετώνται. Το Σέγγεν τώρα. Πολλοί στάθηκαν σε αυτό, όντως είναι ένα σύμβολο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σύμβολα. Δεν μπορώ τώρα να σας πω πολιτικές παρατηρήσεις μια που είμαι υπάλληλο. Θα σας τα πει ο, ο Επίτροπος. Αλλά αυτό το οποίο τώρα μελετούμε είναι πώς θα μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις όχι μονομερός αλλά συνετικά. Γιατί μέχρι σήμερα μπορεί ένα κράτος μέλος να πει στην Κομισιόν και στα άλλα κράτη-μέλη ότι για λόγους ε, εθνικής ασφάλειας αποφασίζει να ξεκινήσει συνοριακούς ελέγχους. Και υπενθυμίζω ότι μια τέτοια απόφαση δεν επιδέχεται δικαστικό έλεγχο. Δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΔΕΚ. Είναι θέμα τελείως διακυβερνητικό. Ο σκοπό είναι να αλλάξουν το σύστημα να έχουμε ένα σύστημα στο οποίο συλλογικά θα λαμβάνεται η απόφαση για το αν συντρέχει ή όχι λόγος ούτως ώστε να ξεκινούν ή να σταματούν προσωρινή έλεγχη. Το ίδιο ισχύει για το σύστημα αξιολόγηση. Τώρα το κάνουμε κάποιε ομάδε εμπειρογνωμών. Συμμετοχή τη Κομισιόν, και θα εξελιχθεί αυτό σε διαδικασία ομοφωνίας διακυβερνητική. Άρα θα προσθεθεί ένα άρθρο, μια διάταξη και, και και αυτόν τον τρόπο να δούμε κατά πόσο θα έχουμε μια κοινοτικοποίηση και των δύο συστημάτων ελέγχων και αξιολόγησης. Από όσα άκουσα που είπατε, αντιλαμβάνομαι ότι το Κοινοβούλιο προβληματίζεται για το τι θα γίνει, αλλά τελικά θέλετε να εγκαταλείψουμε αυτό το σύστημα της μονομερούς ανάληψης ενέργειας. Να δούμε τι θα καταφέρουμε. Πάντως αυτό είναι ο σκοπός μας. Τώρα όσον αφορά το άσυλο, είπαμε ότι στόχος μας είναι το 2012. Αυτό το προβλέπει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Το έχει πει σε ψηλότερο επίπεδο Κοινοβούλιο αλλά και Συμβούλιο. Οπότε, μια που θα γίνει η Σύνοδος του Ιουνίου να το συζητήσει, μπορούμε τώρα να κάνουμε μια πιο ενιαία συνεπή προσέγγιση και όχι κατάτμιση προσπαθειών. Οπότε και μπορούμε να φτάσουμε σε μια δέσμη μέτρων που θα λαμβάνονται υπόψη με διαφοροποιημένα οι ανάγκες οπότε και να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα καταλήξει σε μια πιο ολοκληρωμένη κατάσταση, ένα σύστημα πιο ευρωπαϊκό ας το πούμε το οποίο μπορεί να ισχύσει μέχρι το 2012 και κατά τη γνώμη μας αυτό θα μας βοηθήσει και μας επικρίνουν ότι έτσι από πλευράς διαδικασίας καταργούμε κάποια συστήματα που ισχύουν, κάποιες διαδικασίες. Άρα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ότι το συζητά το Συμβούλιο. Και θα πρέπει επομένως να συνεργαστούν για αυτό το θέμα Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Και είναι σημαντικό ότι και εσείς το συζητείτε. Και επί τη βάση μας των, προτάσεων που θα κατεβάσουμε τον Ιούνιο θα δρομολογηθεί μια διαδικασία ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε εκεί που θέλουμε. Πάντως, οπωσδήποτε, δεν θα πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία σε επίπεδο Συμβουλίου. Δεν είναι τώρα θέμα ούτε Eurodac ούτε μηχανισμού του Δουβλίνου. Είναι εδώ ένα θέμα πολύ πιο γενικότερο. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο πολιτικό. Τώρα όσον αφορά επίσης το κατά πόσον είναι πρακτικά εφικτή η μεθοριακή έλεγχη. Παράδοξο φαίνεται, αλλά γίνεται. Η Γαλλία για κάποιες ώρες έκανε ελέγχους για λόγους δημοσίας τάξης τα τρένα που ερχόντουσαν από την Ιταλία. Γιατί εφοβάτω η Γαλλία το ότι θα έρθουν κάποιοι για να κάνουν κάποια συλλαλητήρια και διαδηλώσει. Φυσικά και αυτό έφερε κάποια κυκλοφορική συμφόρηση. Φανταστείτε να, να γίνει αυτό μεταξύ κάτω χωρών και Γερμανίας. Ναι, εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο καταφύγιο, τελευταία λύση. Γίνεται λοιπόν και έχει συμβεί. Έχει συμβεί ας πούμε ε, για κάποιες μαζικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και σας ε, επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ελέγξει το κατά πόσο έχει υπάρξει όχληση και ανακοίνωση. Δεν επιδέχεται δικαστικό έλεγχο. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και θεωρούμε ότι αυτό είναι η τελευταία λύση μόνο. Δεν είναι ο σκοπός να δημιουργούνται προβλήματα, να διασπάται η νέα αγορά. Θέλουμε να διευκολύνουμε την κυκλοφορία των ανθρώπων. Δεν θέλουμε να την μπλοκάρουμε. Τώρα κατά πόσο είναι σκόρμο να υποβληθεί άλλη πρόταση. Η πρόταση είναι αυτή που είναι. Θα πρέπει να σταθμίσουμε και τα δύο. Και ό,τι χρειαζόμαστε μετανάστες πρέπει να τους μεταχειριζόμαστε με δίκαιο τρόπο. Θα πρέπει από την άλλη μεριά να υπάρχει ασφάλεια. Θα πρέπει να γίνουμε επίσης, ε, να, να, είμαστε καταφύγιο για κάποιους πρόσφυγες και όλα αυτά πρέπει να φοριστούν όχι μονομερός αλλά συλλογικά. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα. Αυτό θέλουμε να στείλουμε σε κοινοβούλιο και συμβούλιο. Και έτσι τελικά να υπάρξει συνένεση πολιτική. Και έτσι να απεμπλέξουμε μια διαδικασία που τώρα έχει μπλοκαριστεί. Επομένως, ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε, όχι να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Να δούμε. Πώς αφορά την επιστολή, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον έχουμε κάποιον... Όταν ε, έχουμε κάποια επιστολή προς αρχηγό κράτους ή κυβερνήσεως, τότε η συνήθις πρακτική είναι η επιστολή να προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Κομισιόν και όχι από τον Επίτροπο. Δεν είναι αυτό ε, προς έκπληξη. Όσον αφορά τώρα την προσωρινή προστασία, πρόκειται για κάτι που το έχει επαναλάβει από αυτή τη θέση η κυρία Μάλμστον. Πρέπει να κρίνεται αν συντρέχουν κάποιες συνθήκες. Επιδιώκουμε τη συνένεση, αλλά το θέμα δεν είναι να μετράμε απλώς το πόσοι συμφωνούν ή όχι, αν υπάρχει πλειοψηφία ή όχι. Θα πρέπει να διαπιστώνουμε αν συντρέχουν κάποιες συνθήκες. Δηλαδή ένα νομοθέτημα, μια οδηγία. Έχουμε, έχουμε κάποιους που δεν μπορούν να επιστρέψουν γιατί υπάρχει αστάθεια, πόλεμος, επομένως. Το αν συντρέχει αυτή η οδηγία είναι ένα θέμα και το εάν το κράτος μπορεί να στείλει πίσω τους πρόσφυγες αυτό είναι άλλο. για τη Μάλτα. Θα πάμε τρεις πιο χώρα, γιατί έχουμε μια μικρή χώρα όπου πάνε λίγοι. Το έχει επαναλάβει η Επίτροπος πολλές φορές. Ότι αυτή η διάταξη, αυτό το, μέσο, το μέτρο δεν έχει εφαρμοστεί. Θα πρέπει όμως να ζυγίσουμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος. ξεκινάμε με προσωρινή προστασία και μπορεί να καταλήξουμε σε μια πάγια ρύθμιση. Αλλά άλλο το άλλο το άλλο. Τώρα, το ποιος κρίνει το τι ισχύει με τη συνθήκη του Σέγγεν είπαμε ότι θα πρέπει να ορίσουμε κάποιες ε, αρχές, κάποιες βάσεις για να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση ανάλογα με το τι θα πει Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Okay, Mr. We thank you for being here. We thank... Ευχαριστώ κύριε Μανσεβίση. σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεσαν τα μέλη και οι πολιτικές ομάδες. Ελπίζουμε ότι οι ανησυχίες οι οποίες εκφράστηκαν έχουν κάποιο νόημα για τις συζητήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν στο Συμβούλιο. Λοιπόν, είδαμε ότι ο υπεύθυνο διευθυντή της εσωτερική ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ παρόν, Έτοιμο να πάρει το λόγο. Τον καλωσορίζω εδώ λοιπόν στο έδρανο του Προεδρείου και θυμίζω ότι ξεκινάμε μια συνεδρίαση από εδώ και πέρα και κλεισμένων των θυρών. Ευχαριστούμε τον κύριο Μανσερβίση, τον χαιρετάμε. Στέφανο.